Καλησπέρα. Με πολύ χαρά σας βλέπω συνάδελφοι και προσκεκλημένοι ομιλητές και λοιποί προσκεκλημένοι σε αυτή τη διήμερη συνάντηση. Θα ήθελα πρώτα να σας εξηγήσω πώς έχει η μερίσια διάταξη και το, τα χρονικά περιθώρια της σημερινής μας συνάντησης θα αφιερώσουμε μία ώρα από τις 3.30 με 4.30 για την Τουρκία, μετά μία ώρα για τις φυλακές στο Λίβανο και τη Συρία από τις 4.30 μέχρι τις 5.30 και μετά η τελευταία ώρα, 5.30 με 6.30, θα, θα είναι αφιερωμένη στο Καζακστάν. Και θα ήθελα να κάνω δύο ανακοινώσεις για, αυτές τις, για τη Συρία και το Λίβανο πρώτα. Θα θυμάστε ότι θελήσαμε να έχουμε μια κοινή ακρόαση για την κατάσταση των φυλακών στην Παλαιστίνη, το Ισραήλ, τη Συρία και, την... και το Λίβανο αλλά δεν μπορέσαμε να το οργανώσουμε αυτό και γι' αυτό με την άδειά σα, συνεννόηση με, με, ακολουθώντας με βάση τις προηγούμενες αποφάσεις οι φυλακές της Παλαιστίνης και του Ισραήλ θα εξεταστούν στη διάρκεια μιας άλλης ακρόασης μόλις μπορέσουμε να την προβλέψουμε στην ημερήσια διάταξη για το Καζακστάν. Πρέπει να σας πω ότι υπήρξε αίτημα από την πρεσβεία του Καζακστάν που μας ζητούσε να αναβάλουμε την ακρόαση λόγω του γεγονότος ότι σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του Καζακστάν, ο κ. Μπάιεφ, επισκέφτεται τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα βρίσκεται αύριο στο Κοινοβούλιο την ώρα που είχαμε προβλέψει την ακρόασή μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Καζακστάν. Πρέπει να σας πω, να σας διαβεβαιώσω ότι ήταν καθαρή σύμπτωση το ότι συμπίπτουν η επίσκεψή του και η ακρόαση. Ε, χρειάστηκε λοιπόν να αποφασίσω, επειδή έχουμε φορτωμένο πρόγραμμα σήμερα και αύριο, να ακολουθήσουμε αυτά που είχαμε αρχικά προβλέψει για να στείλουμε μάλιστα και ένα μήνυμα στο Καζακστάν ότι θεωρούμε ότι η τωρινή Προεδρία του ΟΑΣΕ θα προωθήσει υψηλά πρότυπα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, είχαμε ο πρόεδρος Μπούζεκ το γραφείο του Πρόεδρου Μπούζεκ, επειδή θα συναντηθεί αύριο με τον Πρόεδρο του Καζακστάν, αύριο Τρίτη, αν μπορούσαμε να έχουμε σήμερα τουλάχιστον και όχι αύριο την ακρόαση για το Καζακστάν. Αυτό το δεχθήκαμε, νομίζω ότι ήταν το μόνο ε, που μπορούσαμε να κάνουμε και με τα χαρά καλωσορίζουμε τους εκπροσώπους της πρεσβείας του Καζακστάν εδώ στις Βρυξέλλες στη συνεδρίασή μας γιατί το πρόγραμμα το αυριανό μετά από τον χρόνο των ερωτήσεων η ιδέα είναι να εξετάσουμε την έκθεση εντεκίνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι τις 10.30 κατόπιν θα αφιερώσουμε 10.30 με 10.30 μία ώρα για το Τουρκμενιστάν και τέλος μία ώρα με το διευρυμένο Προεδρείο από τις 11.30 μέχρι τις 12.30. Αυτή λοιπόν είναι η προτινόμενη ημερήσια διάταξη και ερωτώ εάν συμφωνείτε, αν μπορούμε να την εγκρίνουμε. Φαίνεται ότι ναι, εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη και κάποιες ανακοινώσεις. Βραβείο Ζαχάροφ. Ο κύριος Γιγέρμου Φαρίνας επελέγει φέτος για το βραβείο Ζαχάροφ και αποφασίστηκε από την διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου αυτό την περασμένη Πέμπτη. Η τελετή θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου και η Μονάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας καταβάλει προσπάθειες για να οργανώσουμε τον αρτιότερο δυνατό τρόπο αυτή την τελετή. Ελπίζω και εύχομαι ότι ο Πρόεδρος αποφασίσει να καλέσει έναν, ε, τον Όλοφ, έναν από τους περσινούς ε, νικητές του βραβείου Νόμπελ να είναι παρόν, ε, συγγνώμη, να είναι παρόν επίσης. Ο κύριος Όρλοφ αυτή τη στιγμή βρίσκεται ε, έχει, έχουν απαγγελθεί εναντίον του κάποιες ποινικέ κατηγορίες και δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να φύγει από τη χώρα όπως μάθαμε την περασμένη εβδομάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε προηγούμενες περιστάσεις όταν ε, χορηγήθηκε ε, σε, το, το, το βραβείο Ζαχάροφ ορισμένοι αποδέκτες δεν ήταν δυνατόν, είχαν κάποιες δυσκολίες να έρθουν να το παραλάβουν. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν ο Κισολόφ θα μπορέσει να έρθει τελικά το Δεκέμβριο ή αν αποφασίσει, επιλέξει να αφήσει κάποιον άλλο να μιλήσει για λογαριασμό του. Ο πρόεδρος καλεί τις κυρίες με τα λευκά, τις πρώην, ε, στις οποίες είχε απονεμηθεί στο παρελθόν το βραβείο Ζαχάροφ και δεν είχαν τότε τη δυνατότητα να το παραλάβουν. Μόλις έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα θα τις μοιραστούμε βεβαίως με τα μέλη της Επιτροπής. Για τον κύριο Φαρίνια τα τελευταία νέα είναι ότι είναι πολύ αδύναμος αλλά και ετοιμάζεται να ξεκινήσει νέα απεργία πίνης αν δεν του επιτραπεί να ταξιδέψει. Τώρα, δύο λόγια για τη διαδικασία του βραβείου Ζαχάροφ. Ο πρόεδρος εκλήθη ζητήθηκε από τον πρόεδρο να αποφευθούν συγκρούσεις σε ό,τι αφορά την απονομή των βραβείων. Καλούμαστε όλοι να σκεφτούμε το θέμα. Μιλώντας με πολλούς συναδέλφους από διάφορες πολιτικές ομάδες και βλέποντας αυτά που είχαν συζητηθεί στις συνεδριάσεις θα πρότεινα να πούμε ότι η τελική απόφαση για τον βραβείο Ζαχάροφ να γίνει με μυστική ψηφοφορία όλων των Ευρωβουλευτών και με παραπάνω από ένα γύρο ψηφοφορίας εν ανάγκη. Συνομιλώντας με συναδέλφους αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει επιθυμία, μεγάλη επιθυμία να συμμετέχουν όλοι πιο ενεργά στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και αυτό να το συζητήσουμε μεταξύ μας. Σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε μια πιο δίκαιη και πιο δημοκρατική απόφαση. Θα ήθελα να σας θυμίσω για την Ολομέλη της περασμένης εβδομάδας ε, εγκρίθηκαν πολλά σημαντικά ψηφίσματα και όλα αυτά που θα αναφέρω συμμετείχαν ενεργά σε αυτά τα μέλη Ουκρανία, Ζυμπάμπελ, Μολδάβα, Καμπότζη, Ρωσία με συμμετοχή δυναμική όλων των μελών της υποεπιτροπής μας. Το θέμα των διαπραγματεύσεων για τους νέους κανονισμούς για το Ευρωπαϊκό Όργανο Εκδημοκρατισμού και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προχωράει όπως συμφωνήθηκε πέρσι καταρχή, ε, την περασμένη εβδομάδα συγγνώμη, καταρχήν από το Κοινοβούλιο. Με αυτό σημαίνει στην ουσία ότι το Κοινοβούλιο δεν συμφωνεί με τη στάση, τη θέση του Συμβουλίου. Το Συμβουλίο δεν θέλει να δεχθεί αντιπροσώπευση always insist on the inclusion of delegated acts for all decisions fulfilling the criteria. Κατεχώρηση σύμφωνα με το άρθρο το σχετικό άρθρο τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διατηρηθούν οι προνομίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το τομέα. Κύριε Λουμπίλερ, η οποία έχει εργαστεί μαζί με την κυρία Γκάλ για την έκθεση όσον αφορά το μέσο και δημοκρατισμό και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και ελπίζουμε ότι θα ευωδώσουν οι διαπραγματεύσει την ερχόμενη εβδομάδα. Υπάρχει μια δικούσα επιτροπή η οποία παρακολουθεί τις ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και να δούμε πώς θα καταφέρουν να προωθήσουν τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, για μια, δύο λόγια για την ίδρυση της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Την περασμένη εβδομάδα ε, πέρασε η σχετική νομοθεσία και τώρα περιμένουμε τα επόμενα βήματα, τα επόμενα στάδια. Θα ήθελα να ξέρετε ότι πήρα διαβεβαιώσεις από τη Βαρόνια Άστον ότι καμιά απόφαση για τη θέση των, ε, ευρω... ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια της υπηρεσίας έχει... δεν έχει ληφθεί ακόμα Πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε τα σημαντικά μας αιτήματα και την πρόοδό τους ώστε στις δομές να ενταχθούν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υπάρχει μία τμήμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο με στρατηγικές αρμοδιότητες. Θα σημειώσατε ότι υπάρχει στι 3 το απόγευμα την Τετάρτη μια συνεδρία τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου θα είναι παρούσα η εκπρόσωπος, εκπρόσωπο για να συζητήσει μια σειρά από θέματα πολιτική με τα μέλη. Αυτή δεν είναι βεβαίω μια ευκαιρία για να συζητήσουμε για τι οργανωτικέ δομέ, αλλά θα τι θυμίσω στο μέτρο του δυνατού με μια επιστολή η οποία θα ε, περιέχει και θα αναλύει τις αποφάσεις που θα έχουμε λάβει εδώ. Σας λέω επίσης ότι αυτή τη βδομάδα την Πέμπτη εγώ εξ ονόματος όλων μας όλων των μελών της Επιτροπής εκλήθη να λάβω μέρος σε μια άτυπη συνεδρίαση COP η οποία θα οδηγήσει στην ε, εκβάθρον αναθεώρηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι που θα το συζητήσουμε αύριο στο Διευρυμένο Προεδρείο, διότι αυτή είναι μια πολύ χρήσιμη ευκαιρία για όλους μας να παρουσιάσουμε ορισμένες ιδέες και σκέψεις στη συζήτηση με τους ακολούθους για τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατών μελών. Συνάδελφοι, θα ε, σοκαριστήκατε μετά από τις αποκαλύψεις για τις ευθύνες ε, της, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας για κάποιες εκτελέσεις και βασανιστήρια, βασανιστήρια έρευνες πρέπει να ξεκινήσουν σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της ε, των βασανιστήριων. Υπονομεύεται το κύρος των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης σε κάποιο ποσοστό, γι' αυτό πρέπει να παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις αυτών των τομέα. Η, δια... η ο, διάλογος, ο διατλαντικός διάλογος για την νομοθεσία θα επαναληφθεί, θα συμμετέχουν ορισμένοι από εμά και αυτή θα είναι μια πάρα πολύ κατάλληλη ευκαιρία να προωθήσουμε την αποφάσή μας να συνεργαστούμε με μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου για όλα τα θέματα που άπτονται της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είπαμε και το Μάιο στα πλαίσια της αντιπροσωπείας μας που επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον τον Μάιο. Ο αναπληρωτής υπουργό Εξωτερικών του Βιετνάμ, ο κύριος Κβάν Μπιντς Μίτς, ήθελε μια βίντεο διάσκεψη με εμένα εξ ονόματος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με τον κύριο Ρόμπερτ Γκόμπελ, ο οποίο είναι αντιπρόεδρο της ε, αντιπροσωπείας ΑΣΕΑΝ. Ήταν στο, είχαν έρθει στις Βρυξέλλες, εμείς είμαστε στο Στρασβούργο, αλλά είχαμε μία σύνδεση βίντεο με την αντιπροσωπεία του Υπουργού του Βιετνάμ, η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ο λόγος για τον οποίο ήθελε να ανταλλάξει απόψεις μαζί μας ήταν η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ Βιετνάμ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. μπορεί να μην χαιρετήσαμε την υπογραφή αυτής της συμφωνίας τη λάβαμε υπόψη μας και μοιραστήκαμε, μοιραστήκαμε, τη, με τους εκπροσώπους του Βιετνάμ τις ανησυχίες μας για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τους είπαμε ότι έχουμε ψηφίσει ένα ψήφισμα στις 26 Νοεμβρίου 2009 για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ ε, όπου εκφράζουμε μεγάλες ανησυχίες για τα δικαιώματα των σκεφτικών κομμάτων. Και τις πάρα πολύ ε, βαριές ποινές ε, για τους bloggers που φτάνουν μέχρι 11 ε, χρόνια και την δίωξη θρησκευτικών κοινοτήτων όπως η Καθολική Εκκλησία ή τους οπαδούς του βουδικού μοναστηρίου Μπατνάτ. Είχαμε πιστεύω μια χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων και ελπίζω ότι ο Υπουργό αντιλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχει πλέον αρμοδιότητα, πλήρη αρμοδιότητα να πει ναι ή όχι στην υπογραφή διεθνών συμφωνιών. Και ελπίζω συνάδελφοι ότι θα συμφωνήσουμε τι σημαίνει αυτό για την υποεπιτροπή μας όταν συζητήσουμε τις επόμενες διεθνείς συμφωνίες που πρόκειται να υπογραφούν. Ο Υπουργός κατανόησε ότι περιμένουμε πιο θετικά μηνύματα από τις βιετναμικές αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα του βραβείου Νόμπελ, η αντιπροσωπεία στο Πεκίνο μετέφερε τα συγχαρητήρια του Προέδρου Μπαρόσου στη σύζυγο του Λιοξία Πότς, την κυρία Λινξία. Αλλά αυτό που συνέβη ήταν όταν ένας ανώτερος διπλωμάτης πήγε στην κατοικία της κυρίας Λινξία, συνοδευόμενος από διπλωμάτες άλλων χωρών, τους δεν τους επιτράπει από φύλακες η είσοδος. η, η Λούξια δεν έχει τη δυνατότητα να βγει από το σπίτι της, δεν μπορεί να επικοινωνεί με κανένας. Ο άντρας είναι εδώ και παραμένει ακόμα στη φυλακή. Η ποινή του είναι 11 χρόνια. Και μπορώ να σας πω ότι είπατε εκπρόσωπος η κυρία Άστον μέσω της εκπροσώπου της κάλεσε τον τύπο να αντιδράσει σε αυτό το συμβάν και ζήτησε την απελευθέρωση του λιοξίου. Επίσης κάλεσε τις κινέζικες αρχές να θέσουν τέρμα στην ε, κατοίκον κράτηση που έχει επιβληθεί στη σύζυγό του. Τέλος, για την Ουγκάντα. Σε μια από τις χειρότερες εφημερίδες, Rolling Stone είναι ο τίτλος της στην Ουγκάντα, εικόνες και διευθύνσεις πάνω από 100 φιλοφίλων δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, καλώντας τους αναγνώστες να τους βρουν και να τους κρεμάσουν. Τίποτε λιγότερο από αυτό. Εξ ονόματός μας, ελπίζω να μου επιτραπεί να καταδικάσω αυτή τη συμπεριφορά και να καλέσω την κυβέρνηση του της Ουγγάντα να εξασφαλίσει την προστασία, την ασφάλεια αυτών των ατόμων. Καλό επίσης την Παρόνια Άστον, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη να αναλύσουν προσεκτικά την κατάσταση, την κατάσταση στο Ιονουγκάντα ε, για λόγους γενετήσου προσανατολισμού και να προωθήσουν το σεβασμό αυτών των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα θυμάστε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε ένα ψήφισμα για ε, ένα σχέδιο νομοθεσίας κατά το, της ομοφιλοφιλίας στην Ουγγάντα τον περασμένο Δεκέμβριο. Λόγω διεθνών πιέσεων ο νόμος αυτός δεν ψηφίστηκε τελικά. Αλλά παρόλα τα αυτά πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις προσεκτικά σε περίπτωση που δεν αρχίζουν να βελτιώνονται τα πράγματα. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις ε, της Προέδρου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ερχόμαστε τώρα στο θέμα 3 στην ημερήσια διάταξη ακρόαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία εν ώψη της έκθεσης προόδου της Επιτροπής της 9 Νοεμβρίου 2010. Αυτή είναι μια τακτική ετήσια ακρόαση που οργανώνουμε στην υποεπιτροπή μας θα προσπαθήσουμε να σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή στο πλαίσιο της παρακολούθησης ε, της προόδου της Τουρκίας να τηρήσει τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Οι διαπραγματεύσεις ένταξης συνεχίζονται εδώ και πέντε χρόνια. Πάνω από πέντε χρόνια μάλιστα και είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και προς το συμφέρον της Τουρκίας και του τουρκικού λαού να παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις των, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Τα θέματα που θα συζητήσουμε είναι γνωστά σε περισσότερους από εμά, ελευθερία έκφραση, ελευθερία τύπου, ελευθερία, θρησκευτική ελευθερία, κοινωνικά, πολιτιστικά δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων και κακομεταχείριση ε, σε, σε κρατούμενους των από την αστυνομία. Υπάρχει μια σημαντική απόφαση του Ιουνίου 2010 στην Τουρκία, περίπτωση βασανιστήριων. Επιβλήθηκαν σε νέα αξιωματικού αστυνομίου βαρύτατε ποινέ. Και αυτή, αυτό είναι ασφαλώ ένα βήμα προς τα μπρο για την καταπολέμηση της ατιμορρησία κρατικών λειτουργών και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή προσπάθεια. Η γενική εικόνα δεν είναι απόλυτα σαφής. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά δημοσιογράφων, ε, συντακτών, συγγραφέων που δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις ελεύθερα. Μια... Θα ήθελα να αναφέρω την περίπτωση Ντόγκαν Ακανλή, ακτιβιστή, ο οποίος στις 10 Αυγούστου 2010 συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης όταν πήγαινε να ταξιδέψει να δει τον άρρωστο πατέρα του. Φαίνεται ότι κρατείται από τον 20 Αυγούστου 2010 διότι δήθεν ήταν, είχε εμπλακεί σε μια ληστεία του 1999 σε ένα ανταλλακτήριο συναλλάγματος στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά είναι προφανές ότι αυτή η διαδικασία εναντίον του που έχει κινηθεί οφείλεται στο γεγονός ότι μίλησε για τις ε, σφαγές των Αρμενίων και χαρακτηρίζοντας την ως γενοκτονία. Η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα παρακολουθεί τη δική του και την περίπτωση και τις περιπτώσεις άλλων από πολύ κοντά. Τώρα, με πολύ χαρά καλωσορίζω τους προσεκλημένους ομιλητές μας για τη συζήτηση ο κύριος Άντρου Γκάρντνερ πρώτον που είναι ο ερευνητής για την Τουρκία της Amnesty International κατόπιν μια δικηγόρο την κυρία Χούλια Γιούστερση που είναι νομική σύμβουλος του Ιδρύματο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Τουρκίας η οποία ασχολείται ειδικότερα με νομικές υποθέσεις για αντιρρησίες συνείδησης. Κατόπιν η κυρία Αλεχάνδρα Χκάζ Γκράνγκε, διευθυντή για την Κροατία, την, Κροατία, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία, την Τουρκία, την Ισλανδία, από την Γενική Διεύθυνση Διεύρυνση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα καλωσορίζω, κυρία Κασγκράνια. Και θα ήθελα επίση να καλωσορίσω τον πρέσβη, τον κύριο Σελίμ Κούνεραλπ, που είναι ο μόνιμο αντιπρόσωπο τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστούμε κύριε πρέσβη που ήρθατε και Έχουμε δύο συναδέλφους οι οποίοι είναι οι κύριοι εκπρόσωποι μας ε, στα θέματα των σχέσεων με την Τουρκία. Η κυρία Ελεν Φλότρ αφενός, πρόεδρος της αντιπροσωπείας ε, ε, της κοινή κοινοβουλευτική Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και τη κυρία Όμεν Ράιτεν που είναι η συγγήτρια για την Τουρκία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία ελπίζω ότι θα έρθει σύντομα οι παρουσιάσει δεν πρέπει να ξεπεράσουν τα 10 λεπτά. Θα είμαι πολύ αυστηρή μαζί σα αν ξεπεράσετε το χρόνο σα. Και θα καλέσω αμέσω τον κύριο Άντρου Γκάρνερ από την Amnesty International να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λίγες παρατηρήσει μονάχα στη γενική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία για μία σειρά από θέματα όπως είπε, είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει τροποποίησεις νομοθεσία και κάποιες βελτιώσεις στην καθημερινή πρακτική, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, συνεχιζόμενες παραβιάσεις, ενώ συγχρόνως φαίνεται με την ατζέντα για την νομοθετική αλλαγή που είναι επιτάπτω στην Τουρκία, υπάρχουν δυνατότητες για αλλαγές στο άμεσο μέλλον αν εξετάσουμε τις ε, τροποποιήσεις του συντάγματος οι οποίες εγκρίθηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εφόσον υπάρχει πολιτική θέληση. Αλλά βλέποντας επίσης αυτές τις μεταρρυθμίσεις μπορούμε να δούμε ότι ήταν και κάπως και θα μπορούσαν να ήταν πιο αποτελεσματικές αυτές οι μεταρρυθμίσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Εάν εξετάσουμε την κατάσταση των βασανιστήριων και της κακομεταχείρισης στην Τουρκία, εξακολουθεί να ισχύει ότι ω Amnesty International, ως Διεθνής Αμνηστία, παίρνουμε συνέχεια καταγγελίες, αξιόπιστες καταγγελίες για βασανισμούς και κακομεταχείριση σε επίσημους χώρους κράτησης όπως είναι τα σοφρονιστικά καταστήματα και η αστυνομική σταθμή στην Τουρκία αλλά επίσης και κακομεταχείριση εκτός επισήμων χώρων κράτησης κατά τη διάρκεια της ε, ε, μεταγωγής σε αστυνομικούς σταθμούς ή φυλακές και κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. Όλες αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστούν πέραν της κακομεταχείρισης σε επίσημους χώρους κράτησης. Κάτι ακόμα το οποίο είναι σημαντικό Υπάρχει το θέμα της ατιμορρησίας για βασανισμό και κακομεταχείριση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη σοβαρότητα από ό,τι μέχρι τώρα. Εάν η ίδια και κηρυγμένη πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης για μηδενική ανοχή για τα βασανιστήρια πρόκειται να γίνει κάποτε πραγματικά αποτελεσματική. Το θέμα αυτό της ατιμορρησία είναι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσει και η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστήριων όταν εξετάσει τον επόμενο μήνα την έκθεση που αφορά την Τουρκία. Στον τομέα αυτό μπορώ να πω ότι υπήρξαν κάποιες θετικές εξελίξεις, παραδείγματος χάρη η απόφαση στην περίπτωση που αφορούσε την, ε, τον θάνατο του Αγγέν Σαμπάν, ο οποίος πέθανε το 2008 ενώ ήταν σε κράτηση, για πρώτη φορά καταδικάστηκαν κρατικοί αξιωματούχοι για προξένηση βασανιστήριων που οδήγησαν στο θάνατο αυτό όμως εξακολουθεί να είναι ακόμα η εξαίρεση. Η πιο συνηθισμένη κατάσταση είναι ότι δεν υπάρχουν, δεν συνέχεια σε καταγγελίες κατά κρατικών αξιωματούχων και δεν διώκονται για τέτοιες περιπτώσεις βασανιστήριων ή κακομεταχείρισης. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να σταθώ και σε ορισμένε άλλες μεμονωμένες περιπτώσεις που καταδεικνύουν το γενικό κλίμα που επικρατεί στην Τουρκία και ε, όχι τις εξαιρέσεις. Ο, υπήρξε ένας νεαρός ο οποίος πυροβολήθηκε το 2007 με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτος μετά από αυτό το γεγονός αφού τον πυροβολήσαν οι αστυνομικοί υπήρξαν ορισμένες αστοχίες στην ε, ε, έρευνα που έγινε χάθηκαν ουσιώδεις μαρτυρίες, δεν υπήρξε μια έγκαιρη διερεύνηση, υπήρξαν καταγγελίες και απαγγελία κατηγοριών κατά του θύματος και μετά από τρία χρόνια ο Φεργάτ ε, Γκέτσεκ αυτή τη στιγμή είναι υπόδικος και κινδυνεύει να καταδικαστεί σε μεγαλύτερη ποινή από ότι οι αξιωματικοί της αστυνομίας οι οποίοι κατηγορούνται για τους πυροβολισμούς που τον άφησαν παράλληλο. Μια άλλη περίπτωση για την νοτιοανατολική Τουρκία. Ο Ρεσούλ Ιλτσεν πέθανε, έχασε τη ζωή του σε συνθήκες κράτησης πέρσι και η διερεύνηση αυτού του γεγονότος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε από χρόνο λόγος για απαγγελία καταγορίας κατά κρατικών αξιωματούχων παρά το γεγονός ότι ευρέθηκαν σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι και σε άλλα τμήματα του σώματος του ατόμου αυτού. Δεν θα υπάρξει λοιπόν καμία δίωξη που θα ακολουθήσει το θάνατο του υπό συνθήκες κράτησης. Επίσης έχουμε το πρόβλημα των παιδιών τα οποία διώκονται βάσει αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας για την υποτιθέμενη και την καταγγελόμενη συμμετοχή τους σε διαδηλώσεις ενώ έχουν λάβει χώρα τροποποιήσει στην νομοθεσία που δεν επιτρέπουν αυτά τα παιδιά να διώκονται βάσει τη αντιτρομοκρατική νομοθεσία, κάτι το οποίο το χαιρετίζουμε. Υπάρχουν πολλέ καταγγελίε ότι κατά τη διάρκεια τη ε, δίωξη και τη εξέταση αυτών των παιδιών λαμβάνουν χώρα βασανιστήρια και κακομεταχειρήσει, οι οποίε δεν διερευνούνται στη συνέχεια. Έχουμε λοιπόν τέτοιε περιπτώσει για αυτά τα παιδιά τα οποία υφίστανται διώξει και εξάλλου πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν περάσει πολλού μήνε σε κράτηση, σε συνδίκες κράτησης, αλλά δεν υπάρχει καμία προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί η αποκατάστασή τους μετά από την έξοδό τους από τις φυλακές, από την πλευρά των τουρκικών αρχών. Αν εξετάσουμε το θέμα της ελευθερίας έκφρασης επίσης, έχουμε μια κατάσταση όπου υπάρχει μεγαλύτερη τόλμη, τολμούν να εκφράσουν τη γνώμη τους οι δημοσιογράφοι και απλοί πολίτε για θέματα όπω η κατάσταση των Αρμενίων στην Τουρκία και για τα γεγονότα του παρελθόντο. Παράλληλα όμως βλέπουμε να υπάρχει αύξηση ποινικών δικών κατά δημοσιογράφων ή ε, συγγραφέων που είναι αντιφρονούντες προς τις επίσημες απόψεις και ιδίως σε ό,τι αφορά το κουρδικό θέμα είναι περισσότερες οι υποθέσεις στα δικαστήρια που έρχονται και υπάρχει μεγαλύτερη καταφυγή στην αντιτρομοκρατική νομοθεσία η οποία μπορεί να επισύρει αυστηρότερες ποινές από άλλες νομοθετικές διατάξεις. Ενώ λοιπόν γίνεται το δημοκρατικό άνοιγμα στην Τουρκία, οι αντιφρονούντες εξακολουθούν να διώκονται και να τους απαγγέλλονται κατηγορίες βάσει της ε, Αντιτρομοκρατική και άλλη νομοθεσία, και αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να μπορεί κανεί να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του. Επίση, για τους πρόσφυγε και του ετούντε ασύλου υπάρχει εκεί δυνατότητα βελτίωση τη κατάσταση, Αυτή τη στιγμή το καθεστώ κράτηση, το οποίο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεωρήθηκε άνομο, εξακολουθεί να παραμένει. Συνεχίζονται αυτές οι συνθήκες παράνομης κράτησης αλλά υπάρχει τώρα ένα νομοσχέδιο για την παροχή ασύλου, το οποίο θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της κατάστασης των, ε, των προσφύγων και των ετούντων ασύλου. Αλλά χρειάζεται να υπάρξει και διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και να έρθει ε, το ταχύτερο δυνατό ενώπιον της Μεγάλης Τουρκικής Αθνοσυνέλευσης για να μεταφραστεί σε ένα νομοθέτημα. Φαίνεται όμως ότι η κοινωνία των πολιτών δεν θα, δεν θα τύχει διαβούλευσης όπως θα έπρεπε. Επίσης υπάρχει το θέμα των αντιρρησιών συνείδησης για τη στρατιωτική θητεία στην Τουρκία. Εν συντομία ήθελα να σας αναφέρω ότι το δικαίωμα της ε, αντίρρησης συνείδησης το απορρίπτει τελείως η Τουρκία παρά το γεγονός ότι έχει υποχρέωση να δώσει αυτό το δικαίωμα στους πολίτες της. και έχει υπογράψει τη Σύμβαση για τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα, εξακολουθεί να υπάρχει μια κατάσταση όπου αυτοί οι οποίοι είναι αρνησίστρατοι, αυτοί οι οποίοι αρνούνται για λόγους συνείδησης, την χάνουν ή βασανιστήριων σε στρατιωτικές φυλακές και τα άτομα αυτά τα οποία ασκούν το δικαίωμα για την ε, ε, συνείδησης δεν καταδικάζονται, δεν δικάζονται και καταδικάζονται μία φορά, αλλά κατ' επανάληψη έρχονται ενώπιον των δικαστηρίων για ουσιαστικά το ίδιο αδίκημα. Αυτό φυσικά είναι μία παραβίαση του άρθρου 3 του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην περίπτωση Ιλκερ το 2006 και η απόφαση αυτή που ζήτησε από την Τουρκία να αλλάξει νομοθεσία της για να μην υπάρχει κατ' επανάληψη δίωξη αντιρρησιών συνείδησης μέχρι στιγμής δεν έχει εφαρμοστεί από την Τουρκία και παρόλα αυτά είναι υποσυζήτηση ένα νέο νόμο για την στρατιωτική θητεία στην Τουρκία που δεν αναφέρει καθόλου το θέμα τη αντίρρηση συνείδηση. Κάτι το απογοητευτικό επίση το θέμα τη ελεύθερη έκφραση για τα θέματα της αντίρρησης συνείδησης αυτοί οι οποίοι διεκδικούν αυτό το δικαίωμα δημοσίως πολλές φορές υφίστανται δίωξη βάσει του άρθρου 318 του τουρκικού ποινικού κώδικα που ποινικοποιεί και κολλάζει την αποξένωση των πολιτών από το θεσμό της στρατιωτικής θητείας. Και κάποιος ο οποίος κάνει κάτι τέτοιο πολλές φορές υφίσταται πολλαπλές διώξεις. Για το θέμα λοιπόν της αντίρρησης συνείδησης υπάρχει ένα άτομο, η Ινάν Σιουβάτ, ο οποίος είναι υποκράτηση από τον Αύγουστο του 2010 σε, και σε συνθήκες αφέρτης κράτησης από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα λόγω της άρνησής του να εκτελέσει τη στρατιωτική του θητεία και αυτό για λόγους αντίρρησης συνείδησης. Για μένα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι έχουν γίνει μεν αλλαγέ σε νομοθετικό επίπεδο που έχουν τροποποιήσει και έχουν βελτιώσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Αν εξετάσουμε λοιπόν το, τις πιο πρόσφατες συνταγματικές αλλαγές, θα πρέπει όμως να παρακολουθήσουμε και το πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη. Υπάρχει παραγωγικά στο τουρκικό σύνταγμα το άρθρο 90, μια πολύ, με μια πολύ ισχυρή διατύπωση που λέει ότι όταν υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ εθνικού δικαίου και διεθνού δικαίου για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπερέχει το εθνικό δίκαιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν εφαρμόζεται πάντα από τα δικαστήρια. Και υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία έχουν εφαρμοστεί ανεξάρτητοι φορεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλα αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως το προαιρετικό πρωτόκολλο κατά της, των βασανιστήριων έχει υπογραφεί, έχει μονογραφεί το 2005, αλλά δεν έχει κυρωθεί ακόμα. Θα κλείσω λοιπόν σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Όταν κάνετε την προηγούμενη παρουσίασή σας στην υποεπιτροπή μας, ε, σας σταμάτησα απότομα. Ε, για να μην το κάνω λοιπόν και τώρα, ε, δεν, ήθελα μάλλον να το κάνω και τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Γκάρτνερ. Τώρα θα ήθελα να καλέσω την Χούλια Ουσπέτσι για να μας παρουσιάσει το δικό της θέμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω για την ποινικοποίηση της αντίρρησης συνείδησης στην Τουρκία και τις δυνατότητες που δίνει η εθνική νομοθεσία και νομολογία και το διεθνές δίκαιο. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο σύντομη από, την, από τη Σκόπη επαρχικά. Ελπίζω να τα καταφέρω. Το Σύνταγμα της ε, Τουρκίας προστατεύει την ηθική ε, απόφαση των ατόμων δυνάμει του άρθρου 21 ε, και το άρθρο 25 για το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Πέρα από το Σύνταγμα πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει καμία διάταξη στο Σύνταγμα για την υποχρεωτική φυσιολογική θητεία, ούτε καν για τη στρατιωτική θητεία. Το Σύνταγμα ρητά γνωρίζει την ελευθερία τη συνείδηση. Όμω ο ποινικό νόμο και το ποινικό δίκαιο ε, δεν δίνει δυνατότητα να ασκήσει κανεί το συνταγματικό του δικαίωμα ε, και προτάσει το νόμο από το δικαίωμα. Επομένως, ε, θα πρέπει τα άτομα ε, να ασκήσουν τη στρατιωτική τους θητεία και οι αντιρρησίες ε, συνείδησης θεωρούνται στρατιώτες και γι' αυτό ακριβώς δικάζονται από τα στρατιωτικά δικαστήρια με βάση τον στρατιωτικό ποινικό κώδικα. Ε, αντιμετωπίζονται σε άτομα τα οποία ε, ανυπακούν α, κατά, κατά εξακολούθηση. Επίσης, αντιμετωπίζουν την, το φάσμα της φυλάκησης μεταξύ τριών μηνών και ε, δύο χρόνων. Ε, Εξαιτία αυτού του νομοθετήματος, οι οι αντιρρησίε συνείδηση υφίστανται έναν φαύλο ε, δικών και τιμωριών. Ο Τσαλάρ Τουμπού είναι ένα καλό παράδειγμα που δείχνει ε, το πρόβλημα αυτής της διάταξης. Αυτός καταδικάστηκε μία πρώτη φορά, αλλά ξανά καταδικάστηκε λόγω ανυπακοής μεταξύ των της 29ης Απριλίου 2005 και 13ης Φεβρουαρίου 2006. Το δικαστήριο αρνήθηκε να ερευνήσει τους λόγους για την αντίρρηση συνείδησης και οι εισαγγελείς και τα δικαστήρια θεωρούν ότι τα, οι αντισύσεις συνείδησης έχουν σαν σκοπό να αποφύγουν ε, τη στρατική θητεία και ε, δίνουν κίνητρα και σε άλλους ε, στρατιώτες να κάνουν το ίδιο. Ε, οι αντισύσεις συνείδησης ε, για αυτές τις προθέσεις τους αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης μεταξύ 5 και 10 ετών. Επίση, αντιμετωπίζουν ποινικέ και πειθαρχικέ διαδικασίε ω ε, συνέπεια τη πράξη του και μπορεί να υπάρχουν εδώ και διάφορες επιφαντικά ε, στοιχεία ε, στα πλαίσια τη έννοια τη ανυπακοή. Αυτέ οι διαδικασίε καλύπτουν τι πράξει τη ανυπακοή στι μονάδε του στρατού και στι φυλακέ. Οι φυλακισμένοι αντιρσίε συνείδηση συχνά αντιμετωπίζουν και πειθαρχικέ κυρώσει, καθώ και την απαγόρευση γραφή και λήψη γραμμάτων και επιστολών ε, δεν μπορούν να κάνουν ε, ε, τηλέφωνα και αντιμετωπίζουν και το φάσμα τη απομόνωση. Μεταξύ τη 22η Δεκεμβρίου 2006 και 15η Μαου του 2007, ο Χαλίλ Σάβδα ήταν απομονωμένο στο κελί του για 42 μέρε, γιατί αρνήθηκε να ξηρίσει το μουσι του, να φορέσει τη στρατιωτική στολή και να σεβαστεί άλλε στρατιωτικέ προποθέσει. Ε, οι αντιληψίες συνειδήσεις αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο των βασανιστήριων, ε, κα, της κακομεταχείρισης ε, και τον φαύλο κύκλο βέβαια ε, δικών και καταδικών. Ε, Επίση, συχνά πέφτουν θύματα φυσικών επιθέσεων, τους ταπεινώνουν, δεν μπορούν να ζήσουν την καθημερινότητά τους μαζί με τους άλλους φυλακισμένους. παρά το γεγονός, πρέπει να πούμε ότι Πρόκειται για σαφείς παραβιάσεις ε, των διατάξεων περί απαγόρευσης του βασανιστηρίου και της κακομεταχείρισης. Η μεταχείριση του Οσμάν Μουράτ Ούλκε, Μεχμέτ Μπάλ, Μεχμέν Ταρχάν, Χαλίλ Σάβδα και Ενβέρ Αϊντεμίρ δείχνει ότι η μεταχείριση των αντιρρησιών συνείδησης παραβιάζει όχι μόνο την απαγόρευση του, των βασανιστήριων και της κακομεταχείρισης, αλλά και τη διάταξη περί απαγόρευσης της, ε, των διακρίσεων. Ε, επιπλέον, ε, πέρα από τις διώξεις, τιμωρίες και τις κακομεταχειρήσεις, οι αντιρρησίες συνείδησης διώκονται ποινικά και μερικές φορές καταδικάζονται γιατί δηλώνουν τις πεπιθήσεις τους σε άλλους. Θεωρείται ότι με αυτέ τι δηλώσει, ε, όπου δηλώνουν τα προσωπικά τους κίνητρα, οι αντιρρησίες συνείδησης απομακρύνουν το κοινό από την υποχρέωση στρατητικής θητείας. Άλλες δηλώσεις που υποστηρίζουν την αντίρρηση συνείδησης άλλα άτομα με τέτοιες δηλώσεις αντιμετωπίζουν ε, τον ίδιο κίνδυνο. Και οι αντιρρησίε συνείδηση και άλλα άτομα που κάνουν δηλώσει υπέρ αυτών διώκονται και καταδικάζονται με βάση το άρθρο 318 του τουρκικού ποινικού κώδικα. Οι κυρώσει ε, μπορεί να φτάσουν σε ποινή φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια. Η ποινή φυλάκιση είναι μεγαλύτερη αν οι δηλώσει αυτέ δημοσιεύονται ή μεταδίδονται τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά. Ε, Επίσης, όποιοι εκφράζουν τις απόψεις τους ε, για τους αντιρρησίες συνείδησης και αυτοί αντιμετωπίζουν ε, διώξεις. Παραδείγματο χάρη, ένας ε, δημοσιογράφος, ο Μπιλγκούλ Οσμπαρίς, αντιμετώπισε διάφορες αγωγές επειδή δημοσίευσε στην εφημερίδα Ουλκέντι Οσγκούρ Κούσνα μία σειρά από άρθρα για το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης και αντιμετώπισε μία ποινή φυλάξη 21 χρόνια. Ε, τώρα, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα με βάση την εθνική νομοθεσία. Όπως σας είπα, το Σύνταγμα δεν ε, περιλαμβάνει καθόλου περιορισμούς ε, για την έκφραση της αντίρρησης συνείδησης. Τα δικαστήρια και οι πολιτικές αρχές μέχρι στιγμής παραδοσιακά βασίζονται στο άρθρο 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα, ε, ανθρώπινα δικαιώματα που σημαίνει ότι κάθε χώρα μπορεί να οργανώσει όπως θέλει τη στρατιωτική θητεία. Όμως, το άρθρο 4 Αφορά κυρίως τη δουλεία και τα καταναγκαστικά έργα και μόνο μέσα σε αυτό το πλαίσιο αντιμετωπίζει την αντίρρηση συνείδηση. Το Συμβούλιο τη Ευρώπη ε, έχει λάβει αποφάσει που ξεπερνούν αυτέ τι διατάξει ε, του άρθρου αυτού και ζητάει από τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με αυτέ τι αποφάσει. Επιπλέον, το άρθρο 18 τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα, το οποίο επικυρώθηκε από την Τουρκία το 2003, αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων να μην κάνουν την ε, στρατιωτική του θητεία λόγω των απόψεών τους. Είναι αναφυσβήτητο ότι η αντίρρηση συνείδησης θα πρέπει να θεωρείται ως ε, θεμελιώδες δικαίωμα και με βάση το, τις διεθνείς συνθήκες και με βάση το τουρκικό σύνταγμα. Το βασικό θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί είναι η αντισυνταγματικότητα του άρθρου 1 του στρατιωτικού νόμου Μιλάμε για την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και το άρθρο 45 του στρατιωτικού ποινικού κώδικα που ποινικοποιεί την πράξη της αντίρρησης συνήθισης, μια και τα άρθρα αυτά υποσκάπτουν το δικαίωμα που εκφράζω παραπάνω. Η ατυχή συνέπεια της άρνησης αντίρρησης συνείδησης ως δικαίωμα και η απουσία νόμων που να καλύπτουν τις δραστηριότητες των αντιρρησιών συνείδησης είναι ότι οι αντιρρησίες αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν, όπως είπε ο κ. Γκάρνερ, πολλαπλές ε, δίκες. Ο νομοθέτης λέει ότι σε διαφορετικές φάσεις της ε, διαδικασίας ε, σχεδιασμού της νομοθεσίας τα άτομα μπορεί να διαπράξουν διαφορετικά δικήματα. Όμως, μιλάμε για άτομα τα οποία δεν έχουν μια στρατηγική άρνησης. Ε, ο αντιρσίας συνείδησης έχει ένα και μόνο κίνητρο σε όλες τις φάσεις της απόφασής του. Αρνείται να κάνει τη σαδιωτική του θητεία και ό,τι αυτό συνεπάγεται συνολικά. Οι άνωθοι νομικές διατάξεις, σύμφωνα με, με βάση τις οποίες οι αντισίες συνείδησης ε, διώκονται, δεν είναι συμβατές με τις πράξεις τους. Παρά τις αποφάσεις που ε, λαμβάνονται εναντίον του, οι πράξει του όμω δεν έχουν ω πρόθεση τη λιποταξία ή την ανυπακοή. Αντίθετα, όπω δηλώνεται σαφώ από του αντιρρησίε, σε όλε τι φάσει τη διαδικασία έχουν μία και μόνη και αδιάλειπτη πρόθεση και αυτή είναι να αρνηθούν την στατιωτική του θητεία για λόγους συνείδησης και για λόγους ε, πολιτικών πεπιθήσεων. Αυτή η συζήτηση ε, λαμβάνει χώρα και στην Τουρκία και με βάση το τμήμα 5 εγκλήματα του τουρκικού ποινικού δικώδικα και το άρθρο 41.1 ε, κανονικά θα έπρεπε μία ποινή να επιβληθεί αν το ίδιο αδίκημα έχει, έχει διαπραχθεί περισσότερο από μία φορές. Στην περίπτωση όμως του Οσμάν Μουράτ Ούλκε, ε, η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για την αυθαίρετη κράτηση ε, είπε ότι με την καταδίκη του ατόμου αυτού μετά την πρώτη καταδίκη και σύλληψή του ε, η Τουρκία προβαίνει σε παραβίαση της αρχής του Νεμπισινίδεμ. Ε, εξετάζοντας την αίτηση του Οσμάν Μουρά Τούλκε, το, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε ότι οι πολυάριθμες ποινικέ καταδίκες, ε, το σωρευτικό αποτέλεσμα των ποινικών καταδικών, Ε, είχε ε, το δυσανάλογο αποτέλεσμα ε, να οδηγήσει στο να κάνει αυτός ο άνθρωπος τελικά τη στατιωτική του θητεία έμεσα. Αυτές οι διαδικασίες έχουν σαν σκοπό να καταπιέσουν την πνευματική προσωπικότητα του ατόμου, να του εμπνεύσουν το φόβο, το, την, το άγχος, την αίσθηση του ευάλωτου, Στην περίπτωση του Οσμάν Μουράτ Ούλκε, ε, υπάρχει παραβίαση του άρθρου 3 της σύμβασης, γιατί ο άνθρωπος ε, πραγματικά μετά από αυτή την κακομεταχείριση αισθανθόταν με σοβαρούς πόνους ε, και πολλά, είχε πάρα πολλά προβλήματα. Τα άτομα τα οποία διώκονται ε, συστηματικά και καταδικάζονται αντιμετωπίζουν παραβίαση του δικαίωμα τους, του να μην καταδικάζονται, του να μην δικάζονται δύο φορέ ε, και του δικαιώματο στην αντίρρηση, ε, στην αντίρρηση για λόγου συνείδηση. Στι 5 Δεκεμβρίου 2006 συζητήθηκε για πρώτη φορά η υπόθεση Ούλκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ασκήθηκαν ε, και τέθηκαν δύο ερωτήματα. Πρώτον, τα ατομικά μέτρα και τα γενικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν, ούτω ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με την απόφαση του δικαστηρίου ε, για άτομα τα οποία αρνούνται να κάνουν τη στατιωτική του για λόγους συνείδησης ή για θρησκευτικούς λόγους. Θα πρέπει να σταματήσετε. Έχετε ήδη ξεπεράσει τον χρόνο σας. Το 2007 η τουρκική κυβέρνηση ενημέρωσε την Επιτροπή ότι σχεδιάστηκε ένας νόμος ε, και έχει σταλεί στον Πρωθυπουργό. Όμως, ε, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν δίνει στοιχεία για το που έχει φτάσει η διαδικασία. Και μετά το 2007 δεν έχει δοθεί συνέχεια στο νομοσχέδιο αυτό. Το νομοσχέδιο θα πρέπει να προχωρήσει. Θα πρέπει να γίνει από νομοσχέδιο νόμος ούτω ώστε να αναγνωριστεί η αντίρρηση συνείδησης ω ανθρώπινο δικαίωμα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ουστάση για την πλήρη αυτή γνωμοδότηση που δώσατε σε νομικό επίπεδο. Συγγνώμη που σα παρενόχλησα. Σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Πρέπει να κατανοήσετε ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Κάναμε μια ε, εξαίρεση του Γκάρντνερ γιατί τον είχαμε διακόψει την προηγούμενη φορά που είχε λάβει το λόγο ενώπιον μα. Και τώρα βλέπω ότι η κυρία Αλεχάνδρα Κασκάνια είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση. Σας δίνω το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ. Πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ Θα ήθελα να σας πω ποιος είναι ο ρόλος της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Από την Επιτροπή σας και άλλες επιτροπές συχνά δεχόμαστε ατομικές ερωτήσεις για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και οι ερωτώντες μας ε, θέλουν να μάθουν τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να θέσουμε τέρμα σε αυτή την κατάσταση και θα προτερήσω ποιος είναι ο ρόλος της Επιτροπής, τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο ε, λειτουργούμε. Ας ε, επιστρέψουμε στο 99 στο Ελσίνκι. Κρίθη υποψήφια χώρα η Τουρκία, η βάση ήταν σαν αποτέλεσμα είχαμε το 1998 μια πρώτη, με βάση μια πρώτη εκθέση της Επιτροπής την πολιτική οικονομική, οικονομικά κριτήρια και την τήρησή τους από την Τουρκία. Η Τουρκία δεν πληρούσε τα πολιτικά κριτήρια την εποχή εκείνη και ως εκ τούτου απεκλείστη από την έναρξη των προενταξιακών διαπραγματεύσεων. Έκτοτε συνεχίζουμε να δημοσιεύουμε τέτοιες εκθέσεις. Το 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ανοίξει τις διαπραγματεύσεις για ένταξη με την Τουρκία και τον Οκτώβριο 2005 ξεκίνησαν ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις. Η να, ληφθούν, να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στηρίχθηκε σε μια αξιολόγηση ότι η Τουρκία πλέον επαρκώς πληρούσε τα πολιτικά κριτήρια που περιλαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Ε, προηγουμένως δεν πληρούσε επαρκώς τα κριτήρια, τώρα πλέον τα, πληρούσε επαρκώς. Με την έναρξη των διαπραγματεύσεων, η παρακολούθηση της ε, Τουρκίας για την τήρηση των πολιτικών, πολιτικών κριτηρίων συνεχίστηκε. Στο κεφάλαιο 23 περιλαμβάνονται τα ανθρωπίνα δικαιώματα, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά το κεφάλαιο αυτό δεν έχει ακόμα ανοίξει με την Τουρκία. Η Επιτροπή παρουσίασε την έκθεσή της στο Συμβούλιο και η έκθεση εξετάζεται από το Συμβούλιο διότι η αναγκαία ομοφωνία που απαιτείται για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις δεν έχει ακόμα επιτευχθεί σε επίπεδο Συμβουλίου. Παρακολουθούμε λοιπόν τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με, αυτό, με την ετήσια έκθεση προόδου, τις εργασίες των υποεπιτροπών, τις επιτροπές σύνδεσης και τα συμβούλια σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και η διαδικασία, και η διαδικασία των διαπραγματεύσεων εκτός του κεφαλαίου 23 το οποίο ακόμα δεν έχει ανοίξει. Το άρθρο 86 του συνδείξη Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η νομική μας βάση που προβλέπει τα θεμελιώδη δικαιώματα έτσι όπως προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να γίνονται σεβαστά και να και αποτελούν τις θεμελιώ... μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακολουθούμε λοιπόν το νομικό πλαίσιο και την ε, εφαρμογή του. Κάτι που δεν συμβαίνει συχνά πάντοτε στην Τουρκία. Υπάρχουν πάρα πολλά δικαιώματα που αναφέρονται στο χαρτί αλλά δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Ελευθερία του συνεταιρίζεσθε. Ε, και επίσης υπάρχουν ε, ορισμένες ε, περιπτώσεις δίωξης ομοφιλόφιλων και λεσβίων που και αυτές δεν, τηρούν, δεν τηρούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Καταλήγουμε σε συμπεράσματα για κάθε κατηγορία θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση μεμονωμένες περιπτώσεις. Γι' αυτό είναι σημαντική η συνεισφορά μας στην απόψινή ακρόαση τα ευρήματά μας τα υποβάλλουμε, τα θέτουμε υπόψη των τουρκικών αρχών σε όλα τα επίπεδα, σε συνεννόηση μαζί τους. Παρέχουμε επίσης και οικονομικές ενισχύσεις σε πολιτικά όργανα στην Τουρκία προσπαθώντας να, τους κάνουμε, να, τα κάνουμε, να κάνουμε τα μέλη τους να αντιληφθούν πώς πρέπει να εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν για την ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεστε, του συνεταιρίζεσαι κλπ έτσι όπως ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζουμε θερμά τις ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών με 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ώστε να ενισχύονται και να υποστηρίζονται δραστηριότητες αυτών των οργανώσεων και να τους βοηθήσουμε να ενισχύσουν το δίκτυό τους. Τώρα, θα ήθελα να μιλήσω για την κατάσταση σήμερα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. 12 χρόνια παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία έχουν συμπληρωθεί. Και όλα αυτά αναφέρονται στις αιτήσει εκθέσεις πρόοδου. Όταν προετοιμάστηκα για αυτή την ε, ακρόαση, εξέτασα όλες, μελέτησα τις προηγούμενες εκθέσεις πρόοδου και ειδικότερα τα κεφάλαια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το φετινό, ε, η φετινή έκθεση θα δημοσιευθεί σύντομα και βλέπουμε από τις εκθέσεις πρόοδου 98 μέχρι 2010 ότι έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος αλλά υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν στην Τουρκία. Μέχρι το 2003 οι ετήσιες εκθέσεις μας υπογράμμιζαν ότι η θανατική ποινή εξακολουθούσε να περιλαμβάνεται στον ποινικό κώδικα και περιγράφουν τη συνεχιζόμενη συζήτηση για την κατάργησή τη στην Τουρκία. Το 2004 μπορέσαμε να ανακοινώσουμε ότι η θανατική ποινή επιτέλους είχε καταργηθεί. Θα ήθελα να αναφερθώ και στο θέμα της σημερινής συζήτησης το νομικό, νομοθετικό πλαίσιο της Τουρκίας δεν ρυθμίζει επαρκώς το θέμα των αντιρρησίων συζήτησης. Εκείνο που αρνούνται να κάνουν στατιωτική θητεία για ε, λόγους συνείδησης ή θρησκευτικού λόγους αντιμετωπίζουν ε, αυστηρές κυρώσεις και ποινές. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε μια απόφαση του 2006 στην περίπτωση σε μια υπόθεση ότι αυτή η συμπεριφορά παραβιάζει το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της να εφαρμόζει ε, το, το, διατάξεις του άρθρου και να εκτελεί τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Τουρκία. Το 1998 είχαμε γράψει στην ετήσια έκθεσή μα ότι επαναλαμβανόμενε περιπτώσει εξαφανίσεων, εξοδικαστικών εκτελέσεων και βασανιστήριων συνεχίζονταν. Τα πράγματα έχουν ευτυχώ αλλάξει προς το καλύτερο έκτοτε. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει προσπάθεια συμμόρφωσης με ορισμένες ε, βασικές νομοθετικές διατάξεις αλλά παρόλα τα αυτά υπάρχουν ακόμα και πάρα πολλές παραβιάσεις για την ελευθερία έκφρασης. Πριν από 12 χρόνια είχαμε γράψει ότι μια πολύ στενή ερμηνεία του συντάγματος και άλλων νομοθετικών διατάξεων χρησιμοποιείται για να επιβάλλονται ποινές σε συνδικαλιστές, συγγραφείς, μέλη ΜΚΟ κλπ. για δηλώσεις, για απόψεις που εκφράζουν, για άρθρα που δημοσιεύουν, κάτι που θα γινόταν απόλυτα αποδεκτό σε άλλα, στα κράτη της Ευρώπης, σε άλλα κράτη, στα κράτη της Ευρώπης. Τώρα έχουν γίνει ορισμένες αλλαγές στα, άρθρα του τα σχετικά άρθρα του ποινικού κώδικα και αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα μια εκτεταμένη συζήτηση για αυτό το θέμα στην Τουρκία. Ωστόσο, ο τουρκικός νόμος δεν εγγυάται παρκώς την ελευθερία της έκφρασης. Οι δημοσιογράφοι υφίστανται διώξεις και δίκες ακόμα επειδή έχουν παραβιάσει την αρχή της εμπιστευτικότητας μια συνεχιζόμενη δικαστική διαδικασία. παρόλο που οι πληροφορίες που κομίζουν είναι ήδη ε, δημόσια διαθέσιμες. Τιμωρούνται εάν ε, αναφέρονται στο κουρδικό υπάρχουν απαγορεύσεις λειτουργίας ιστοσελίδων που είναι υπερβολικά δυσανάλογες. Ο τύπος υποχρεώνεται να είναι φιδωλός σε αυτά τα οποία αναφέρει στις δημοσιεύσεις του. Και η Τουρκία βρίσκεται στην 138η θέση στην σημερινή κατάταξη, σε πολύ πιο χαμηλά από ό,τι στο παρελθόν, λόγω επανειλημμένων παραβιάσεων των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων. Ε, θρησκευτική ελευθερία. Στο, στο, στο, χαιρετήσαμε τον εορτασμό που έγινε στην Παναγία Φουμελά, αλλά θα απαιτηθούν σε αυτό το τομέα πάρα πολλές ακόμα προσπάθειες. Έχει γίνει κάποια πρόοδος για την, ε, την ε, ε, επιστροφή ιδιοκτησιών σε θρησκευτικού οργανισμούς, μοναστήρια κλπ. Αλλά τα θρησκευτικά, οι θρησκευτικές οργανώσεις δεν έχουν νομική προσωπικότητα, νομική ιδιότητα δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα οι σχετικέ ε, συνομιλίε. ανθρώπινα δικαιώματα. Το 1998 γράψαμε ότι δεν υπήρχαν ειδικέ διατάξει για την καταπολέμηση τη ε, βία κατά των γυναικών στο γάμο, στον αστικό κώδικα. Πλέον σήμερα ε, υπάρχει σχετική διάταξη μετά από αλλαγή του συντάγματος αλλά θα χρειαστεί να γίνουν προσπάθειες ώστε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο να μετατραπεί, να μετατραπεί σε πραγματικότητα. Διότι εξακολουθούν ακόμα να υπάρχουν προβλήματα με τους υποχρεωτικούς γάμους και την ενδοοικογενειακή βία. Τώρα, η αντιτρομοκρατική νομοθεσία πρέπει επίσης να μεταβληθεί για να μην περιορίζει υπερβολικά την άσκηση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν ε, ε, ε, εκπληρωθεί ορισμένες προσδοκίες σε αυτό το τομέα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο τα τελευταία 12 χρόνια στην Τουρκία με αποτέλεσμα να αρχίσουν και οι διαπραγματεύσεις για ένταξη. Αλλά έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι πολλά χρειάζεται ακόμα να γίνουν διότι όλο και νέες περιπτώσεις, μεμονωμένες περιπτώσεις έρχονται περιπέτουν στην αντίληψή μας με αποτέλεσμα να διαπιστώνουμε ότι δεν τηρούνται πλήρως τα κριτήρια που έχουμε θέσει. Πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τα πολιτικά κριτήρια η Τουρκία για να εδραιώσει η δημοκρατία που θα στηρίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο κράτος δικαίου στη χώρα. Οπωσδήποτε έχουν γίνει κάποια, έχουν γίνει, έχει γίνει μια αρχή αλλά μια αρχή σε μια, σε μια διαδικασία συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων που όμως δεν ολοκληρώνονται ποτέ πλήρως. Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι σε 9 Νοεμβρίου η Επιτροπή θα εκδώσει την έκθεση ε, του 2010, η οποία θα υποβληθεί από τον Επίτροπό μα, τον Επιτροπούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ πληροφοριακά αυτά που μας είπατε. Μας δώσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα οπτική γωνία για όλα αυτά τα οποία έχουν επιτευχθεί τα τελευταία 12 χρόνια και τι παραμένει ακόμα να γίνει. Και τώρα με μεγάλη χαρά δίνω το λόγο στον πρεσβευτή κύριο Σελίμ Κούνεραλ. Ο, είναι ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με αδειμονία περιμένουμε τις αντιδράσεις σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά είμαι εδώ ενώπιόν σα και έχω την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις για τις μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία και ιδίω σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις των τελευταίων 11 μηνών από τότε που είχαμε την τελευταία ανταλλαγή απόψεων. Χαιρετίζω αυτή την ευκαιρία γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παίζει και σημαντικό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Θα ήθελα καταρχήν να υπογραμμίσω μερικά βασικά γεγονότα στη διαδικασία μεταρρύθμισης της Τουρκίας και να απαριθμίσω κάποιες από τις σημαντικές αλλαγές που έχουν γίνει. Οι αλλαγέ που έγιναν σε νομοθετικό επίπεδο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την εδραίωση τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία τη διαδικασία ένταξη τη Τουρκία και επομένω μια υψηλή προτεραιότητα για την Τουρκία. Αλλά είναι απαραίτητε αυτέ οι αλλαγέ για να εκπληρωθούν οι του τουρκικού λαού για περισσότερη δημοκρατία και μεγαλύτερο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από το 2001 η Τουρκία έχει προχωρήσει σε μια εκτεταμένη διαδικασία μεταρρυθμίσεων που συμπεριέλαβε τρει σημαντικέ τροποποιήσει του συντάγματο και επίση ένα νέο αστικό και ποινικό κώδικα, ενώ συνεχιζόταν αγώνα κατά τη τρομοκρατία ω τμήμα τη διαδικασία αυτή της μια από τι πιο σημαντικέ τροποποίησεις του συντάγματο αφορά το άρθρο 90 μετά από την τροποποίησή του το 2004 οι διεθνείς συμφωνίες σε περίπτωση σύγκρουση με το εθνικό νόμο υπερέχουν του εθνικού νόμου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό ευθυγραμμίζει την νομοθεσία στα ευρωπαϊκά πρότυπα σε ό,τι αφορά την ελευθερία έκφραση συγκεκριμένα και έχει μειωθεί σημαντικό αριθμό διώξεων μετά από την έγκριση αυτή τη νομοθεσία. Ο νέο νόμο περί ιδρυμάτων βελτιώνει πολύ την κατάσταση των ε, ε, διεθνών δραστηριοτήτων των Ιδρυμάτων του επιτρέπει επίση να έχουν και οικονομική υποστήριξη και άλλε χορηγίε. Για τον αγώνα κατά της ε, και των βασανιστήριων ήταν θέμα προτεραιότητα, Η πολιτική μηδενική ανοχής όπως τονίσατε και εσεί η ίδια κυρία Πρόεδρε προχωρά και θέλω να χαιρετήσω αυτά που είπατε το θέμα. Έρχομαι τώρα στις πρόσθετες, στις πρόσφατες μάλλον συνταγματικές αλλαγές που είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα στη διαδικασία μεταρρύθμισης και τις ε, εξελίξεις που έχουν λάβει η χώρα το τελευταίο χρόνο. Το πακέτο συνταγματικής μεταρρύθμισης έγινε βάσει των κριτηρίων της Κοπεχάλης και τροποποιεί πάνω από 20 άρθρα του τουρκικού συντάγματος εδραιώντας τις αρχές του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της ε, νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΕΔΑΔ και αντίστοιχε άλλε αρχέ. Με το πακέτο αυτό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδει ελευθερίες έχουν διευρυνθεί, όπω αναγνωρίστηκε από πολλού αμερόληπτους παρατηρητές μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ των βελτιώσεων λοιπόν που έχουν επέλθει είναι η συμπερίληψη της θετικής διάκρισης ως συνταγματικού δικαιώματος για γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και ανάπηρους, επίσης συνταγματικές εγγύησεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων και επίσης σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών και προστασία τους, διεύρυνση της ελευθερίας του συνέρχεστε και συνεταιρίζεστε, άρση των περιορισμών για το ταξίδι στο εξωτερικό, δημιουργία διοικητικού επιτρόπου, ε, δυνατότητα δικαστικού ελέγχου για τις αποφάσεις του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ε, δυνατότητα προσφυγής κατά αποφάσεων δημοσίων υπαλλήλων, το δικαίωμα μεμονωμένης προσφυγής στο Συνταγματικό Δικαστήριο, τροποποίηση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και της λειτουργίας του και επίσης τροποποίηση, μεταρρύθμιση του Ανώτατου Δικαστηρίου Εισαγγελέων και Δικαστών και μια ακόμα σημαντική αλλαγή ήταν η συνταγματική εγγύηση ότι δεν μπορούν πλέον οι πολίτες να δικάζονται από στρατιωτικά δικαστήρια. Μετά λοιπόν από την έγκριση αυτού του πακέτου, το Κοινοβούλιο της Τουρκίας θα δώσει την πρώτη προτεραιότητα στην εφαρμογή αυτού του πακέτου και την ε, υλοποίησή του σε νομοθετικό επίπεδο. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω κάποιες άλλες νέε ιδέε, όπω παραδείγματο η δημιουργία ενό εθνικού φορέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενό θεσμικού φορέα και επίση ενό φορέα κατά τη διάκριση και υπέρ τη ισότητα ανδρών και γυναικών, που επίκειται η δημιουργία του επίση. Για τα δικαιώματα των γυναικών. Εξακολουθεί να είναι προτεραιότητά μα. Η ισότητα των φύλων ενώπιον του νόμου είναι συνταγματική αρχή και οι φόνοι τιμή κολλάζονται με πιο αυστηρές ποινές από το νέο ποινικό κώδικα μέχρι και ισόβια ποινά, μέχρι και ισόβια δεσμά. Ε, επίσης, μετά από την εφαρμογή του κοινού προγράμματος για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ε, γυναικών και των, και κοριτσιών, ε, με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών σε έξι επαρχίες της Τουρκίας από το 2006-2009, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει μια εγκύκλιο ώστε να προωθηθεί μια σειρά από πρωτοβουλίε για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών. Για την θρησκευτική ελευθερία υπήρξε μια εγκύκλειος που εκδόθηκε το Μάιο του 2010 από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες από όλες τις θρησκευτικές κοινότητες είναι αναπόσπαστο τμήμα του τουρκικού έθνους και η προστασία του δικαιώματος θρησκευτικής ελευθερίας για τι θρησκευτικέ μειονότητε δεν είναι μονάχα νομική επιταγή, αλλά έχει και μεγάλη σημασία για να μπορούν να νιώθουν ότι είναι πράγματι όλοι αυτοί τμήμα του τουρκικού έθνους και κράτους. Στις 15 Αυγούστου του 2010, για πρώτη φορά μετά από το 1993, έγινε μια θρησκευτική τελετή στην Παναγία Σουμελά, κοντά στην Τραπεζούντα, με την παρουσία Ορθοδόξων χριστιανών από όλο τον κόσμο και μια αντίστοιχη τελετή έγινε στην εκκλησία του Ακταμά στη Λιμτούβάν, τον Σεπτέμβριο του 2010. Αυτή η αρμενική εκκλησία είχε ήδη ανακαινιστεί και ανοίξει ως μουσείο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού το 2007. Έγινε για πρώτη φορά εκεί μια θρησκευτική τελετή μετά από 95 χρόνια με παρουσία πάνω από 4.000 ατόμων και ε, εγκαταστάθηκε και ο Σταυρός πάνω στην, ε, στον τρούλο της Εκκλησίας στην αρχή αυτού του μήνα. Ένα άλλο θέμα είναι τα δικαιώματα των παιδιών. Το 2010 ενεκρίθη μια τροποποίηση του νόμου κατά της τρομοκρατίας που εξασφαλίζει ότι όλα τα, όλοι οι ανήλικοι, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θα αντιμετωπίζονται από τα δικαστήρια ανηλίκων με τον ίδιο τρόπο. και δεν θα υπάρχει ανάκριση ε, ανηλίκων χωρίς την παρουσία δικηγόρου. Έχουν, είναι υποχρεωτική λοιπόν η νομική τους προστασία. Θα υπάρχει και υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους και τα δικαστήρια ανηλίκων θα γίνονται πάντα, θα λαμβάνουν χώρα και κλεισμένων των θυρών και έχει απαγορευτεί η χρήση χειροπεδών για τους ανήλικους. Επίσης, για τη χρήση άλλων γλωσσών εκτός από τα τουρκικά στα μέσα ενημέρωσης και στη τηλεόραση. Ο νέος κανονισμός για τις εκπομπές επιτρέπει να χρησιμοποιούνται άλλες γλώσσες και διάλεκτοι από Τούρκους πολίτες. Αυτό εγκρίθηκε από το Ανώτατο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο στις 19 Νοεμβρίου 2009 και έτσι έχουν αρθεί όλες οι μορφές περιορισμού για τη χρήση αυτών των γλωσσών και όλες οι νέες αιτήσει για δημιουργία σταθμών έχουν εγκριθεί. Υπάρχουν 15 εθνικοί σταθμοί, 9 τοπικές τηλεοράσεις κτλ. που ε, έχουν το δικαίωμα να εκπέμπουν, να έχει εγκριθεί να εκπέμπουν στις διαλέκτους Ζάζα και Κορμαντζή των Κουρδικών. Προτού ε, κλείσω, θέλω να επανέλθω στο θέμα των ε, αντιρρησιών συνείδησης, το οποίο είναι το ιδιαίτερο θέμα μας σήμερα, και θα ήθελα να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει αποφασίσει ότι είναι δικαίωμα η αντίρρηση συνείδηση βάσει του, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απλώς είπε το, Ευρωπαϊ... το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ότι η Τουρκία δεν έχει επιτύχει να εφαρμόσει πλήρως τις υποχρεώσεις της σε σχέση με την αποφυγή ε, εξευτελιστικής και επάνθρωπης μεταχείρισης. Αλλά η απόφαση του ΕΔΑΔ δεν έδωσε δεν εδραίωσε δικαίωμα σε αντίρρηση συνείδησης, όπως και όλες οι άλλες αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα ληφθεί υπόψη από την τουρκική κυβέρνηση και είναι επίσης σαφές ότι λόγω της συνέχισης της τρομοκρατικής βίας στην ε, Τουρκία είναι περιορισμένο το περιθώριο ελιγμών των τουρκικών αρχών στον τομέα αυτό. Έχουν λίγα ακόμα δευτερότητα. Θα ήθελα να τονίσω ότι η έγκριση της νομοθεσίας βέβαια δεν είναι κάτι που ταυτίζεται με την εφαρμογή της ίδιας νομοθεσίας. Εμείς αποδίδουμε ίση σημασία και στην έγκριση νομοθεσίας και στην εφαρμογή της και γι' αυτό έχουν ξεκινήσει σημαντικά προγράμματα για να εξασφαλιστεί η εκπαίδευση των μελών των δυνάμεων ασφαλείας και των δικαστικών αρχών. Μία ακόμα πρόταση, αν μου επιτρέπετε. Βέβαια, έδωσα απλώ ένα αδρό περίγραμμα των μεταρρυθμίσεων που έχουν λάβει η χώρα στην Τουρκία μέσα στο τελευταίο χρόνο αλλά θα ήθελα να κλείσω υπενθυμίζοντάς σας ότι το μεγαλύτερο ότι η ευρεία πλειοψηφία που υποστήριξε την ε, συνταγματική αλλαγή το Σεπτέμβριο του 2010 καταδεικνύει τη θέληση του τουρκικού λαού να προχωρήσει προς την κατεύθυνση και της ελευθερίας και της δημοκρατίας ακριβώς δηλαδή τις αρχές που συμμεριζόμαστε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορώ μονάχα να εκφράσω την ελπίδα τους επόμενους μήνες όταν εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έκθεση για την Τουρκία θα ενθαρρυνθεί το τουρκικό έθνος να συνεχίσει την πρόοδό του και την ε, προετοιμασία του για να γίνει πλήρως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρέσβη. Σας ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε προς αυτήν την κατεύθυνση και το μήνυμα αυτή τη συνταγματική μεταρρύθμισης είναι προφανώς θετικό. Την επόμενη εβδομάδα, μάλιστα, θα πάω με την πολιτική μου εβδομάδα στην ε, Κωνσταντινούπολη και θα συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Τώρα, μετά τους ε, ομιλητές, τους εξωτερικούς και τον πρέσβη, μπορούμε να περάσουμε στους ευρωβουλευτές. Ε, το λόγο έχει πρώτα η πρώην πρόεδρος αυτής της υποεπιτροπής. θα έλεγα πέντε λεφτά ο καθένας για να έχουμε και χρόνο για τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Γιατί αν μιλήσετε περισσότερο δεν θα υπάρχει χρόνος για συζήτηση. Και νομίζω ότι δεν το θέλει κανένας αυτό. Ε, να ξεκινήσουμε λοιπόν με την κυρία Ελέν Φλότχα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σε πέντε λεφτά δεν μπορώ να σας κάνω μια έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά να σας μιλήσω για, λιγάκι για την κατάσταση του δημοκρατισμού, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, θέματα πιο πολιτικά, το θέμα των Κούρδων, το νέο σύνταγμα ή και τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην Τουρκία είναι ένα ζήτημα επίμαχο που ταλανίζει την κοινωνία και τους πολιτικούς αλλά και τις οργανώσεις ε, και την κοινωνία των πολιτών. Το 2009, παραδείγματο χάρη, ε, είχαμε 12 καταδίκες της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, στα πλαίσια της ελευθερίας έκφρασης. Μία διαβόητη περίπτωση, δυστυχώς πολύ διάσημη, ήταν η δολοφονία ενός ατόμου που είχε για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των δικαίωσε ρήμην, ε, αποφάσισε ότι όχι μόνο η ελευθερία έκφρασή του είχε παρεμποδιστεί, αλλά και το τουρκικό κράτο δεν είχε προβεί στα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του ανθρώπου αυτού. Είναι μια κεφαλαίου σημασία απόφαση και πολύ σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση και το τουρκικό κράτος αποφάσισε να μην κάνει α, έφεση εναντίον αυτής της απόφασης του δικαστηρίου. Δηλαδή τελικά οι τουρκικές αρχές σήμερα αναγνωρίζουν και δεσμεύονται να εφαρμόσουν τα συμπεράσματα των αποφάσεων αυτών του δικαστηρίου, τουλάχιστον στα πλαίσια της περίπτωσης Χραντίνγκ. Τώρα, για την ατιμορρησία των δημοσίων υπαλλήλων. 35 διαδικασίες ε, αγωγές έχουν ε, ξεκινήσει που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν ε, τις ε, πρακτικές πάνω από 400 δημοσίων υπαλλήλων. Η αρμόδια επιτροπή του τουρκικού κοινοβουλίου η ίδια ε, εκφράζει θλίψεις για το λόγο ότι καμία από αυτές τις διαδικασίες δεν οδήγησε σε καταδίκη κάποιου δημοσίου υπαλλήλου. Βλέπετε λοιπόν τις ζημώσεις που γίνονται στον πολιτικό χώρο, στην ε, τουρκική κοινωνία. Και αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Γιατί μόνο τότε θα συνειδητοποιήσουμε και τις δικές μας ευθύνες ως Ευρωπαίοι πολίτες ε, για τη δημοκρατία στην Τουρκία. Νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές ε, καταδίκες είναι λίγο αντιφατικές και παράδοξες. Είναι παράδοξο το, κάτι το οποίο λέμε συνέχεια που είναι κάποια πρότυπα, ε, κάποιες ελευθερίες, η ελευθερία έκφρασης, ε, του συνέρχεστε άνδρων και γυναικών, ισότητα άνδρων και γυναικών και παράλληλα τα κεφάλαια τα οποία θα μας, μπορούσαν να μας επιτρέψουν σημαντικές προόδους, ε, δικαιοσύνη, εσωτερικές υποθέσεις, τα κεφάλαια αυτά για πολιτικούς λόγους μπλοκάρονται, για να μην πω μικροπολιτικούς λόγους. Είμαστε κοινοβούλοι εδώ και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τις ευθύνες μας απέναντι σε αυτό το θέμα. Το τελευταίο που θέλω να πω. Η υιοθέτηση του πακέτου για το Σύνταγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το περιεχόμενο είναι σημαντικό αυτή τη μεταρρύθμιση του Συντάγματο. Αλλά και γιατί το πακέτο αυτό ε, υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρκικό πληθυσμό. Τι σημαίνει αυτό. Σήμερα οι αρχές, για να μην πω και το σύνολο των φορέων ε, και φορέων και εμπλεκομένων στην ε, Τουρκία έχουν σήμερα το πολιτικό περιθώριο να κάνουν μια δουλειά για ένα νέο σύνταγμα. Το νέο αυτό σύνταγμα θα επέτρεπε να θέσουμε το κουρδικό πρόβλημα με τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Σήμερα στον Διαρμπακύρη έχουμε 150 ακτιβιστές που δικάζονται με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Αυτός ο νόμος δεν έχει αλλάξει όπως υπόθηκε. Επίσης υπάρχουν πάντα ανήλικοι για αυτούς τους λόγους ε, στις φυλακές. Επίσης το κουρδικό επιβάλλει μια αλλαγή της αντίληψης για τον πολίτη και την, το ρόλο του πολίτη. Εξού και η ανάγκη για αλλαγή του συντάγματος. Αυτή την έκκληση την κάνουν πάρα πολλοί πολιτικοί. Αυτή την έκκληση την έκανα και εγώ και πολλοί άλλοι πολιτικοί. Και πολλοί Τούρκοι πολιτικοί ε, είναι υπέρ της ε, διαδικασίας για ένα νέο σύνταγμα που θα μας οδηγήσει σε πραγματική ρήξη με το σημερινό σύνταγμα που είναι προϊόν της Χούντας του 1980. Και θα είναι ένα σύνταγμα συνενετικό ε, όλων των φορέων της κοινωνίας. Είναι απόλυτα εκ των ονουκάνευ αν θέλουμε να υπάρξουν πραγματικά θετικές προοπτικές. Και για όλα τα προβλήματα τα οποία ακούσαμε από τους ομιλητές. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικές οι παρατηρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό ε, και έχει να κάνει με αυτά που υπόθηκαν από προηγούμενους ομιλητές για το μπλοκάρισμα του κεφαλαίου 23. Λοιπόν, η συγκέντρια για την Τουρκία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία. Είναι σημαντική για όλους μας και για τον εισηγητή, την εισηγήτρια που θα γράψει μια νέα έκθεση τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου και σας υπόσχομαι ότι θα μεταφέρω τα συμπεράσματα, θα πάρω μαζί μου τα συμπεράσματα αυτής της ακρόασης και θα συμπεριληφθούν στην επόμενη έκθεση. Αυτό που θα ήθελα να πω επίσης είναι ότι εκτιμώ ιδιαίτερα την ενημέρωση ε, για τα πολιτικά θέματα. Πολύ καλή, λέω στη γραμματεία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ουσιαστικό στοιχείο των κριτηρίων της Κοπενχάγης. Τα κριτήρια της Κοπενχάγης για μένα είναι πιο σημαντικά από το άνοιγμα και το κλείσιμο κεφαλαίων. Ας το πούμε αυτό, ξεκινώντας. Η πρόοδος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία συνεχίζεται, αλλά τα τελευταία χρόνια, το είπαν, το είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές και ο πρέσβης, ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα, ψηφίστηκε νέα νομοθεσία Ωστόσο, ωστόσο η πραγματικότητα δεν ακολουθεί πάντα αυτά τα οποία περιέχονται στην νομοθεσία, διότι η εφαρμογή αυτή της νομοθεσία είναι συχνά ανεπαρκής. Και όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με τη μεγάλη πόλωση που υπάρχει στη χώρα. Η πόλωση δεν αφορά μόνο την πολιτική, αλλά και το δικαστικό, το, το τομέα της δικαιοσύνης και την κοινωνία στο σύνολό της. Και ε, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο από αυτό που γίνεται τώρα. Και θα έρθω σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Πρώτον, η τροποποίηση του συντάγματος Όντως πρόκειται για καλή σημαντική πρόοδο. Αλλά οι τροπολογίες αυτές πρέπει να μεταφραστούν σε νομοθετικές προτάσεις και να εφαρμοστούν κατόπιν. Και θα ήθελα αυτή η διαδικασία να επιταχυνθεί. Δεύτερον, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, θα ήθελα να, προτι... να πω ότι ένα νέο σύνταγμα είναι αναγκαίο για τον εξυγχρονισμό της Τουρκίας. Το δημοκρατικό άνοιγμα που ανακοινώθηκε πέρσι ήταν καλό. αλλά δεν ε, προσέφερε τίποτε το ουσιαστικά καινούριο για τους Κούρδους. Στα νέες τροπολογίες της νομοθεσίας η θέση των παιδιών έχει ασφαλώς βελτιωθεί, δεν υφίστανται πλέον δίωξη, αλλά θέλουμε νέες προτάσεις σχετικά με τα δημοκρατικά ανοίγματα για το κουρδικό η Ευρώπη ήταν πάντοτε, ήταν, έδειξε, πάντοτε αλληλεγγύη ε, για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Και θα ήθελα, θα ήθελα όμως να ζητήσω από την κυβέρνηση αλλά και από την αντιπολίτευση πριν από τις εκλογές να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για αυτό το δημοκρατικά άνοιγμα προς τους Κούρδους. Διότι αν θέλετε μια βιώσιμη λύση είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να γίνει. Θρησκευτικέ ελευθερίες. Πέρσι οργανώθηκαν κάποια σεμινάρια, όπως είπε ο πρέσβης, λειτουργίες σε συμβολικούς χώρους. Αυτά είναι σημαντικά αλλά δεν μπορούμε να χαράξουμε πολιτική επικαλούμενη νέα σύμβολα. Απλώς χρειάζονται συγκεκριμένες δράσεις στην Τουρκία ώστε κάθε θρησκευτική μειονότητα να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα τα οποία πρέπει να είναι εγγυημένα. Και χρειάζονται γι' αυτό συγκεκριμένα βήματα στα πλαίσια του δημοκρατικού ανοίγματο. εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια μετά την εφαρμογή, τη θέσπιση του, της νομοθεσίας για τα Ιδρύματα. Η νομοθεσία υπάρχει, αλλά η εφαρμογή υστερεί. και εξαρτάται για ποια περιοχή μιλάμε, την Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα ή κάποια άλλη περιοχή. Αυτό που μας προβληματίζει είναι η ελευθερία του τύπου και η ελευθερία γνώμης. Ορισμένα άρθρα του ποινικού κώδικα εξακολουθούν να εφαρμόζονται, να χρησιμοποιούνται για την δίωξη ε, πολιτών και δημοσιογράφων στο διαδίκτυο πάνω από, άκουσα ότι ε, ε, έκλεισαν πάνω από 6.000 ιστοσελίδε. και αυτό δεν ταιριάζει, δεν ταιριάζει σε μια σύγχρονη δυναμική κοινωνία όπως θέλει να είναι η τουρκική κοινωνία και σε αυτό το τομέα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Μεγάλες, μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί ανήκουν σε σημαντικούς ομίλους που χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ για να προωθήσουν τα οικονομικά τους συμφέροντα. Και σε αυτό, για αυτό το θέμα πρέπει να ψηφιστεί νέα νομοθεσία. Τον περασμένο Μάιο δέχθηκα μια ομάδα δημοσιογράφων και συνδικαλιστών και εκείνοι ζήτησαν μεταρρύθμιση τι νομοθεσίε που αφορά το διαδίκτυο και τα ΜΜΕ. Ο πρόεδρος Γκιούλ την περασμένη εβδομάδα μετά από τη δημοσίευση του World Press Freedom Index παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ανεπάρκειες θέματα που δεν καλύπτονται ακόμα επαρκώς στην Τουρκία. Το τελευταίο σημείο αφορά την Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι αποφάσεις του καθυστερούν εκδίδονται με καθυστέρηση αλλά λίγο πολύ εφαρμόζονται, εφαρμόζονται στην Τουρκία, από την Τουρκία και αυτό οπωσδήποτε είναι ένα θετικό βήμα. Ευχαριστώ για τις πολύ σαφείς παρατηρήσεις σας και για την ε, υπόσχεσή σας να λάβετε υπόψη σας κάποια από τα συμπεράσματα της ακρόασης. Η συζήτηση συνεχίζεται, να σας το υπενθυμίζω. Υπάρχει ενώπιόν μας η έκθεση, η Επιτροπή Ιστορικών Υποθέσεων θα την ε, συζητήσει επίσης. Σας κάνω έκκληση οι πέντε συνάδελφοι που ζήτησαν το λόγο, γιατί έχουμε και το Καζακστάν ακόμα, έχουμε τις φυλακές στη Συρία και το Λίβανο, έχουμε πολλά θέματα. Σας παρακαλώ ε, να περιοριστούν και να μιλήσουν μόνο για ένα λεπτό. Ε, ούτως ώστε να ακούσουμε και κάποιες απαντήσεις. Κύριε Νίλσεν, Γκόσμες, ε, η κυρία Γιαννάκου, Η κυρία Λοχ Μπίλερ είναι η πρώτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σταθώ σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα για τους πολιτικούς ε, κρατούμενους σε φυλακές υψηλής ασφαλείας, ιδίως τον Διερμπακύρ. Ε, για τον κύριο Γκάρνερ είναι η ερώτηση, αλλά και για τους υπόλοιπους ομιλητές, τους οποίους ευχαριστώ για τις γνώσεις τους και την ωραία τους παρουσίαση. Μία ερώτηση. Από ό,τι ξέρω, η κατάσταση στην φυλακή ασφαλείας του Διερμπακήρ είναι προβληματική από άποψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συμφωνείτε με την εκτίμηση αυτή και προς την κυρία Κάσ Κράντζη από την Επιτροπή που είπε ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε ατομικές περιπτώσεις. Μου έφτασε μία επιστολή από ένα κρατούμενο από αυτή την φυλακή υψή της ασφαλείας που είναι πολύ άρρωστος και ο γιατρός του λέει ότι θα ζήσει πάνω από έξι μήνες. οι αρχές ε, μου είπε ότι δεν του επέτρεψαν να πάει σε γιατρό εκτός φυλακής. Ε, ο Υπουργό Δικαιοσύνη ή η Κομισιόν έχει εξετάσει αυτήν την περίπτωση. Η... Αυτό είναι καταδικασμένο σε ισόβια δεσμά. Ε, παρά την καταδίκη σε ισοβια δεσμα παρα μπορεί να αποφυλακιστεί και να πάει στο σπίτι του να πεθάνει τουλάχιστον ελεύθερο. Ευχαριστώ, κυρία Κιλ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τη δημοκρατία θα να μιλήσω, για την καθολική ψηφοφορία. Στο σημερινό πλαίσιο που ανέφεραν οι συνάδελφοί μου, οι δίκες στο Διερμπακύρ και το γεγονός ότι πολλοί δήμαρχοι και αιρετοί άρχοντες ε, σέρνονται ενώπιον δικαστηρίων, ορισμένοι φυλακίζονται και εγώ γνωρίζω το δήμαρχο του Διερμπακύρ, γιατί είμαι από τη Ρέν στη Βρετάνη, που έχει δεσμού συνεργασίες με την πόλη του Διερμπακύρα το 1977. Έχουμε κάποια προγράμματα συνεργασίας αποκεντρωμένα. Γνωρίζουμε αυτή την πόλη λοιπόν και τους, ε, τους αρχοντές τους και το δήμαρχο, το γνωρίζω προσωπικά. Και δεν πιστεύω ότι είναι τρομοκράτη. Είμαι κατάπληκτη. Ε, όταν θελήσαμε να τον φιλοξενήσουμε, α, του είπαν ήδη από τον Ιανουάριο ότι αποκλείεται να μπορέσει να φύγει από την Τουρκία. Κύριε Πρέσβη, μιλήσατε για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Κατά την άποψή σα, είναι εύκολα τώρα. Ο Δήμαρχο όμω του Διαρμπακύρ δεν μπόρεσε να ταξιδέψει. Στην περιοχή μου ε, μιλάμε τα Βρετόνικα. Έτσι. Δεν καταλαβαίνουμε πώ οι Κούρδοι δεν μπορούν να μιλήσουν τη γλώσσα του. Το, το θέμα αυτό τέθηκε και στη δίκη αυτή. Γιατί οι κατηγορούμενοι θέλησαν να μιλήσουν κουρδικά κατά τη διάρκεια τη δίκη του. Η τελευταία μου ερώτηση. Πώ θεωρείτε ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση στο κουρδικό χωρίς να δεχτείτε να συνομιλήσετε με τα άτομα αυτά, τα οποία είναι ενώπιον του δικαστηρίου. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση λύσης χωρίς την συμμετοχή αυτών των ανθρώπων που έχουν εκλεγεί δημοκρατικά από το λαό της περιοχής. Σα παρακαλώ, θα είμαι λίγο πιο αυστηρή με το χρόνο ομιλία. Ε, είχατε φτάσει ήδη στα δύο λεφτά, κύριε Γκόμε. Συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν από τους προλαλήσαντες, την κυρία Φλότχα, την κυρία Ερμαν Ρόιτε. Εμείς είμαστε Ευρωπαίοι και έχουμε ευθύνε. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα κριτήρια της Κοπενχάγης γίνονται σεβαστά. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν γιατί το κεφάλαιο 23 για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει μπλοκαριστεί είναι από τα μπλοκαρισμένα εμπασπιτώσει κεφάλαια. Θέλω επίσης να συμφωνήσω με αυτό που υπόθηκε για τη σημασία του συνταγματικού πακέτου. Αλλά το οποίο δεν είναι παρκές για να αντιμετωπίσει το κουρδικό πρόβλημα, το οποίο είναι κεφαλαίο του σημασίας. Θα ήθελα να πω επίσης ότι παρά κάποιες προσπάθειες προς σωστή κατεύθυνση, ότι υπάρχει μία έτσι πολύ έξυπνη καταστολή ειδικά σε ποινικέ διαδικασίες ε, που το αντικείμενό του η ελευθερία έκφρασης κτλ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Τούρκο πρέσβη. Οι, του, οι στρατιωτικοί δεν εξακολουθούν, οι Τούρκοι στρατιωτικοί να παίζουν ένα υπερβολικά υψηλό και σημαντικό ρόλο. Και εγώ είμαι Πορτογαλίδα και χρειάστηκε να πείσουμε τους στρατιωτικούς για να πάνε πίσω στα στρατόπεδά τους και να αφήσουν το κράτος να λειτουργήσει δημοκρατικά μετά την ε, ε, δικτατορία, για την ατιμορρησία. Θα λογοδοτήσετε για τη συνεργασία σας ε, στις έκτακτες αυτές απαγωγές και κρατήσεις. Κυρία Γιαννάκου, σας παρακαλώ πολύ σύντομα, γιατί δεν θα ακούσουμε καθόλου ε, απαντήσεις. Πολύ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη. Oh, good. Eh, eh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε. Και η κυρία Νίλσεν και η κυρία Γκόμες μίλησαν για το θέμα των Κούρδων και το θέμα της γλωσσικής σου έκφρασης. Ο κύριος Πρεσβευτής αναφέρθηκε σε κάποιες διαλέκτους στην Τουρκία. Όχι, ναι, δεν είναι διάλεκτη, είναι γλώσσες ενός πληθυσμού με μακρά ιστορία, 14 εκατομμύρια τουλάχιστον. Εγώ βρίσκω σκανδαλώδες ότι δεν υπήρξε καμία πρόοδος η οποία έχει επιτευχθεί για τη χρήση της γλώσσας αυτής. Δεν θα επανέλθω στα θέματα των δικών που έχουν γίνει στην περίπτωση του Χραντίνγκ. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το θέμα των βασανιστήριων Είπατε ότι υπήρξε εκεί μια βελτίωση, αλλά μήπως είδατε την έκθεση του Μάρτεν Ντούτσερ, ενός Γερμανού ακτιβιστή από τη Γερμανία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που τόνισε ότι έχουν γίνει και γίνονται ακόμα κάθε μέρα στρατιωτικές επιθέσεις κατά του άμαχου κουρδικού πληθυσμού και έχουν λάβει χώρα 20 εξοδικαστικές εκτελέσεις. Έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά όπλα εναντίον του πληθυσμού και έχουν υπάρξει ακροτηριασμοί μετά τη φώνευση ανθρώπων και έχει δώσει και φωτογραφίες στη δημοσιότητα που τα καταδεικνύουν αυτά. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι ο νόμος ε, στηρίζει την ισότητα των δύο φύλων. Όμως η ισότητα για τις γυναίκες έχει σχέση με την οτροπία και τις αντιλήψεις που υπάρχουν. Ποιες είναι οι ενέργειες τις οποίες έχει προβεί το τουρκικό κράτος ώστε οι αντιλήψεις αυτές να διαφοροποιηθούν. Και από την άλλη πλευρά όταν η ηγεσία της χώρας η οποία βεβαίως έχει προωθήσει ορισμένες αλλαγές με το συμβολισμό της μαντήλας δείχνει κάτι διαφορετικό πώς μπορεί κανείς να σκεφτεί για μια πραγματική ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Τι κάνει για τις γυναίκες το κράτος Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γιαννάκου. Εγώ προτείνω να ακούσουμε τον ε, κύριο Πεσβευτή και τους άλλους προσκεκλημένους ομιλητές, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω ε, πάνω από ένα μισή λεπτό τον καθένα. Κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Φλότοχα και την κυρία Ούμεν Ρόιτεν για τις δηλώσεις τους που έχουν πολλά θετικά στοιχεία. Να σταθώ τώρα στα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν, όπως τα έχω καταγράψει. Υπήρξε ένα ερώτημα καταρχήν για ένα τερματικά ασθενή κρατούμενο στο Διάρμπακε. Δεν μπορώ βέβαια να αναφερθώ σε μια περίπτωση την οποία δεν τη γνωρίζω. Βέβαια ο πρόεδρος της Τουρκίας έχει το δικαίωμα να απονείμει χάρη σε ασθενεί οι οποίοι βρίσκονται σε τερματικό στάδιο σε ό,τι αφορά την κατάσταση τη υγείας του και είμαι σίγουρο ότι θα εξεταστεί προσεκτικά και αυτή η περίπτωση. Νομίζω ότι υπήρξε μια παρεξήγηση για την απαγόρευση τη Κουρδική. Δεν υπάρχει κουρδική γλώσσα η οποία ήταν υπό απαγόρευση ή κάποια άτομα που δεν είχαν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την κουρδική γλώσσα. Σα είπα ότι υπάρχουν ραδιοσταθμοί και σταθμοί τηλεόραση σε αυξανόμενου αριθμού που χρησιμοποιούν τη γλώσσα αυτή. Ίσως υπήρξε κάποια παρεξήγηση εδώ. Κανείς δεν διώκεται για την χρήση της κουλικής απλώς και μόνο για συνεργασία με, ε, σε, με τρομοκρατικές ε, οργανώσεις. Υπήρξε αυτή η έκθεση του κ. Μάρτιν Ντούτσερ. Έχω δει τις φωτογραφίες που έχει η έκθεσή του και έχω μία δήλωση εδώ από το νοσοκομείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε σαν πηγή για αυτή την έκθεση που απορρίπτει απόλυτα όλα αυτά, που αρνείται απόλυτα αυτά τα οποία καταγγέλει ο κύριος ε, Ντούτσα. Και θα διανύμω λοιπόν αυτή την ε, έκθεση, θα τη δώσω στο μέσο της γραμματείας σε όλους τους παρόντες. Δεν υπάρχει καμία διάκριση σε επίπεδο φύλων από την νομοθεσία, αλλά φυσικά αυτό συμβαίνει παντού. Το θέμα είναι η εκπαίδευση και η ενσωμάτωση αυτών των νομοθετικών διατάξεων και το Κοινοβουλίο μας έχει δημιουργήσει μια επιτροπή που εξετάζει τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω ευχαριστήσω και την κυρία Ουστέρτση. Δεν νομίζω ότι υπήρξαν κάποια ερωτήματα σε εσά, προς εσάς. Θα επανέλθω στην Επιτροπή. Εμείς έχουμε εξετάσει την κατάσταση στις φυλακές. Έχουμε μια ομάδα ε, ε, αξιολόγησης από ομοτήμους που θα δημοσιευθεί τον Ιανουάριο του 2011. Συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να κυκλοφορούσουν, να δουν την κατάσταση στις διάφορες φυλακές της Τουρκίας και να καταλήξουν σε συμπεράσματα τις οποίες ε, συζητούμε με τις τουρκικές αρχές στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου. Λοιπόν, η περίπτωση που αναφέρατε θα εξεταστεί και θα προσπαθήσουμε να αποκομίσουμε περισσότερες πληροφορίες. Αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω τώρα θα ήταν να δώσω ένα γενικό σχόλιο για όλα τα άλλα ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί. Βλέπουμε στην Τουρκία να υπάρχει μια μεγάλη ένταση. Δεν είμαστε ακόμα σε μια κατάσταση που να έχουμε ένα ισόπεδο γήπεδο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Αυτό που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει στην Τουρκία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, εξακολουθούν όλα αυτά. Θα πρέπει εν καιρό να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα θέματα, αλλά αυτό αποτελεί και μια από τι μεγαλύτερε υποκλήσει που πρέπει να αντιμετωπίσει η τουρκική κοινωνία. Υπήρξε και το θέμα για το κεφάλαιο 23. Μήπω και άλλε χώρε εκτό Γερμανία και Γαλλία μπλοκάρουν αυτό το κεφάλαιο. Προ το παρόν νομίζω όχι, αλλά σίγουρα η ομοφωνία απαιτείται για την, το άνοιγμα αυτού του κεφαλίου. Ξέρετε λοιπόν ποιοι είναι αντίθετοι σε κάθε χρονική στιγμή. Τώρα, αν υπάρξει μια ψηφοφορία, κανεί δεν ξέρει ποιο υποκρύπτεται πίσω από αυτού που έχουν αρνητική άποψη. Πρέπει να πω ότι εδώ χρειάζεται και περισσότερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτέ τι αδιαφανεί δομέ λήψη απόφαση του Συμβουλίου. Είναι πραγματικά απαράδεκτο να μην ξέρουν οι ψηφοφόροι μα τι γίνεται στου διαδρόμου και στο παρασκήνιο. Για τον Άντριου Γκάρτνερ τώρα νομίζω ότι υπήρξαν κάποια ερωτήματα και προ εσά. Ναι, θέλω να απαντήσω στο ερώτημα το οποίο απευθύνθηκε σε μένα για την κατάσταση των φυλακών στον Διάρμπακερ. Νομίζω το πιο σημαντικό που πρέπει να πω είναι ότι όπως και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών η Amnesty International δεν έχει πρόσβαση στους χώρους κράτησης στην Τουρκία γιατί η Τουρκία δεν έχει ε, επικυρώσει το πρόσθετο πρωτόκολλο για την σύμβαση κατά των βασανιστήριων. Επομένω, δεν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθηση των κέντρων κράτηση στην Τουρκία, κάτι το οποίο για μένα είναι απαραίτητο για να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση των φυλακών και των κέντρων κράτηση στην Τουρκία. Φυσικά είχαμε επαφέ και συνεντεύξει με πρώην κρατούμενου και με δικηγόρου οι οποίοι είχαν πρόσβαση στου πελάτε του στι φυλακέ αυτέ και όλα αυτά μα έχουν οδηγήσει πραγματικά σε ανησυχίε σε σχέση με τι φυλακέ υψηλή ασφαλεία σε όλη την Τουρκία, όχι μόνο στο Διάρμπακερ και ιδίως σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ενώσεων στην Τουρκία και του γεγονότος ότι οι κρατούμενοι οι οποίοι θεωρούνται πολιτικοί κρατούμενοι δεν μπορούν να έχουν κοινέ δράσεις και το συνεταιρίζεστε με άλλους κρατούμενους και η εγκύκλειος που έχει εκδοθεί για το ότι οι κρατούμενοι θα πρέπει να έχουν επαφή τουλάχιστον 10 ωρών μέχρι την εβδομάδα με άλλους κρατούμενους. Αυτό δεν εφαρμόζεται σε όλη, την, σε όλη τη χώρα. Σε ορισμένε περιπτώσεις μονάχα μία ώρα τη βδομάδα έχουν το δικαίωμα να αυλίζονται, να συναυλίζονται με τους άλλους κρατούμενους, οι πολιτικοί κρατούμενοι και κατά άλλα είναι απόλυτα απομονωμένοι. Επίσης, ό,τι αφορά την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, υπήρξε ένα ερώτημα το οποίο ετέθη η Amnesty International, έχει τονίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Ιατρικής, που είναι το αρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων δεν έχει ανεξάρτητο χαρακτήρα λόγω της δομής του και γιατί υπόκειται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και αυτό θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να αποκτήσει αυτονομία για να μπορεί να παρακολουθεί τα θέματα αυτά και αυτό το έχει τονίσει και το ε, Συμβούλιο Επιθεωρητών ε, του Προέδρου της Τουρκίας που κατέληξε σε ένα αντίστοιχο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υπάρξει να εξασφαλιστεί η αυτονομία του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής Ιατρικής. Ευχαριστώ τον κύριο Γκάρνερ και όλους σας για τη ε, συμμετοχή σας ε, στη συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί. Αν ε, δεν είχαν ξεπεράσει το χρόνο τους όλοι οι μιλητές, θα είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο με συμμετοχή και άλλων ε, συμμετεχόντων. Αλλά ξέρω ότι αυτό θα επαναληφθεί και την άλλη φορά θα έπρεπε να υπάρχουν σαφείς γραπτέ οδηγίε προ του ομιλητέ, πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει σα ευχαριστούμε για τι πολύτιμε πληροφορίε που μα δώσατε και όπω είπαμε η συζήτηση θα συνεχιστεί. Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο θέμα και στην ημερήσια διάταξη που είναι η κατάσταση φυλακές τη Συρίας και του Λιβάνου. Μπορείτε παρακαλώ να αποχωρήσετε ήρεμα και ήσυχα από την αίθουσα. Και δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω γιατί θα συζητήσουμε την κατάσταση των φυλακών στη Συρία και το Λίβανο. Αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποιες περιπτώσεις στη Συρία, τις οποίες παρατηρούμε με ιδιαίτερη προσοχή, του κυρίου Χάιτε Μαλμάλι, που είναι δικηγόρος 80 ετών, που αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και που βρίσκεται σε φυλακή για ψευδείς πληροφορίες που ενδεχομένως παραβιάζουν το εθνικό αίσθημα. Μπορείτε τουλάχιστον να σταματήσετε να συνομιλείτε μεταξύ σας. Δεν μπορώ να σας ε, εμποδίσω να φύγετε, αλλά μπορώ να σας ε, απαγορεύσω να μιλάτε μεταξύ σας. Πήρε το βραβείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, από την Ελβετία και ήταν και υποψήφιος μου για το βραβείο Ζαχάροφ. Ένας μεταξύ των εννέα που είχαν προταθεί ως υποψήφιοι. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η δική του περίπτωση θα προκαλέσει το ενδιαφέρον όλων και υπάρχει και ο κύριος Μουχάμενταλ Αλχασάνη ο οποίος και αυτός φυλακίζεται ε, βρίσκεται στη φυλακή για το έργο του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Συρία είναι μια χώρα που προσπαθεί να συσφίξει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να εξετάσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Συρία και θα καλέσουμε τον κύριο Νάντιμ Χούρι να πάρει το λόγο και μετά τον κύριο Ήλιας Ελμάλη που είναι ο γιος του Ελμάλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλετε να καλύψω τώρα το Λίβανο ή θα έχω τη δυνατότητα να ξαναπάρω τον λόγο αργότερα. Θα είναι καλύτερο να συζητήσουμε για τις δύο χώρες σε συνδυασμό. Θα αρχίσω με το Λίβανο και θα ολοκληρώσω με τη Συρία ονομάζομαι Ναντίμ Χούρι, με ο επικεφαλής ερευνητής της Human Rights Watch για τη Συρία και το Λίβανο, με έδρα στη Βηρητό. Ευχαριστώ που με καλέσετε εδώ. Θα ξεκινήσω με το Λίβανο, τη συνθήκη στη φυλακή. Υπάρχουν 20 φυλακές στο Λίβανο, η σημαντικότερη είναι η κεντρική φυλακή. Τρία σοβαρά θέματα αντιμετωπίζουμε στο Λίβανο. Και έχουμε πολλές πληροφορίες, διότι το καλό με το Λίβανο είναι ότι παρόλο που είναι κακές συνθήκες στη φυλακή, η πρόσβαση αυτές είναι ε, εύκολη. Είναι λοιπόν εύκολο να αποκτήσει κανείς συστηματικά πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές. Το βασικό πρόβλημα στο Λίβανο είναι ο υπερπληθισμός, ο υπερπληθισμός στις φυλακές το κράτος λέει ότι υπάρχουν, θέσεις για 3.700 ενώ ουσιαστικά οι κρατούμενοι ξεπερνούν τους 5.500. Το πρόβλημα δεν είναι βεβαίως, το θέμα δεν είναι να χτίσουμε πιο μεγάλες φυλακές. Το πρόβλημα είναι η μακρά κράτηση, ο μακρύς χρόνος κράτησης πριν από τη δίκη 66% το συνολικού αριθμού των φυλακισμένων είναι κρατούμενοι ε, υπόδικοι και υπάρχει και η κράτηση ε, ε, και το θέμα της αντιμετώπισης των ξένων κρατουμένων μετά την αποφυλάκησή τους. εκατό των κρατουμένων είναι αλλοδαποί οι οποίοι εκτίουν την ποινή τους. Γιατί αυτοί οι αλλοδαποί βρίσκονται στη φυλακή ενώ έχουν εκτίσει την ποινή τους σε μεγάλ, τόσους μεγάλους αριθμούς. Ο βασικός λόγος είναι σύμφωνα με τη μια εγκύκλη του 2004 η οποία κατά κάποιο τρόπο έχει αναφέρει στο χαρτί την πρακτική που εφαρμόζεται, οποιοδήποτε έχει εκτίσει την ποινή του παραπέμπεται στη Σουρτέ γενεράλ που είναι γενική ασφάλεια, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με του αλλοδαπού. Αυτή η διαδικασία, η παραπομπή σε αυτή την υπηρεσία μπορεί να κρατήσει μήνες και πολλές φορές και παραπάνω από ένα χρόνο. Αυτοί οι αλλοδαποί παραμένουν στη φυλακή δεν έχουν τη δυνατότητα να ε, αντιδράσουν για τη συνέχιση της κράτησής τους. Και υπάρχει το πρόβλημα των προσφύγων και των ετούντων άσυλων. Όταν, ολοκληρωθεί, όταν τελειώσει η εκτίσουν την ποινή του, η Σουρτέ Γενερά του λέει θα σα βάλουμε σαν αεροπλάνο, θα στείλουμε πίσω. Λένε όχι. Τότε ο Λίβανο λέει δεν σα βάλουμε παρά τη θέλησή σα σε ένα αεροπλάνο, θα σα κρατήσουμε ε, στη φυλακή. Και μετά από ε, ένα διάστημα ε, τα άτομα αυτά ε, εθελοντικά, εθελοντικά δέχονται την πρόταση. Αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα. Τώρα, οι συνθήκες, οι ίδιες στις φυλακές. Οπωσδήποτε υπάρχει έλλειψη ε, αερισμού και φωτός. Οι γιατροί του κόσμου σε μια μελέτη που έκαναν ανέφεραν ότι υπήρχε έλλειψη φυσικού αερισμού σε πολλές φυλακές έλλειψη φωτισμού, φωτός στα κελιά σε 13 από τις 20 φυλακές. Οι καταστάσεις υγιεινής είναι πολύ παλιές, βρώμικα λουτρά, βρώμικα αποχωρητήρια. Οι τοπικές ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε 15 από τις φυλακές δεν έχουν κρεβάτια οι κρατούμενοι κοιμούνται σε στρώματα πάνω στο δάπεδο και δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ υποδίκων και καταδίκων. Η τροφή είναι πάντα πρόβλημα. Όσοι έχουν οικογένειες, οι κρατούμενοι που ζουν κοντά, ε, οι οικογένειές τους τους φέρουν φαγητό. Οι αλλοδαποί χωρίς κάποιο, κάποια οικογένεια υποφέρουν. Επίσης, τι συμβαίνει σε περίπτωση έκτακτη ανάγκη. Μετά τις 5 οι φυλακέ δεν μπορούν να ανοίξουν τα κελιά χωρίς την άδεια του εισαγγελέα. Και αυτό σημαίνει καθυστερήσεις με θανατηφόρες συνέπειες πολλές φορές. Στο χαρτί οι δικαστές έχουν το δικαίωμα να επισκέφτονται τα κελιά και να βλέπουν τι συμβαίνει εκεί. Βλέπουν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι δικαστές δεν κάνουν καν τον κόπο κακομεταχείριση και βασανιστήρια. Αυτό δυστυχώς παραμένει μεγάλο πρόβλημα στο Λίβανο στους χώρους κράτησης περισσότερο, στα κρατητήρια και όχι στις φυλακές, αλλά έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις σε φυλακές. Αλλά το, στους χώρους κράτησης κυρίως εφαρμόζονται τα βασανιστήρια και η κακομεταχείριση. Υπάρχει μια φυλακή του Υπουργείου Άμυνας από το 1995 θεωρείται ε, ε, φυλακή, τώρα χρησιμοποιείται σαν χώρος ε, ανακρίσεων και σαν φυλακή. Οι ΜΚΟ δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή τη φυλακή. Η μόνη οργάνωση που έχει πρόσβαση είναι η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού και επειδή, και επειδή δεν δημοσιεύονται οι εκθέσεις της, δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Ο Human Rights Watch και άλλες ομάδες έχουν συγκεντρώσει στοιχεία για βασανιστήρια στη διάρκεια ανακρίσεων, κυρίως για άτομα που θεωρούνται ότι θεωρούνται ε, ύποπτα για κατασκοπία. Αυτά είναι πρόσφατα παραδείγματα τα οποία έχουμε συγκεντρώσει. Μια δεύτερη ε, φυλακή είναι η φυλακή Ρούμιε, η κεντρική και στην οποία η υπηρεσία πληροφοριών έχει καταλάβει ένα μέρος του κτηρίου και υπάρχει και η εγκατάσταση κράτησης αλλοδαπών κάτω από μια γέφυρα σε ένα χώρο στάθμευσης και εκεί οι συνθήκες ε, χαρακτηρίζονται ως άθλιες. Οι λιβανικές αρχές έχουν καταβάλει προσπάθειες για να βελτιώσουν τις συνθήκες στις φυλακές. Υπάρχει ευρεία συζήτηση και παραδοχή ότι αυτή είναι μια κατάσταση ε, που δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί. Προσπάθησαν κάπως να βελτιώσουν τα πράγματα με μια νέα φυλακή για άνδρες του Ζάχλη που άνοιξε τον Απρίλιο φέτος Επίσης προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τον υπερπληθυσμό των φυλακών, συνέστησαν επιτροπές για να μελετήσουν το πρόβλημα. Όταν απελήθη ο πρώτος κρατούμενος τον, ε, Απρίλιο φέτος, ε, αυτό ήταν κάτι το θετικό, αλλά η Επιτροπή η αρμόδια λειτουργεί με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς και τέλος υπάρχει και ένα πενταετές πρόγραμμα σε συνεργασία με μια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά της δικαιοδοσίας για τις φυλακές από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπάρχουν κάποιες πρόοδοι αλλά τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει σημαντικό ρόλο μέσα από τα θεσμικά της όργανα ή μέσα από τα κράτη-μέλη της. Ένα παράδειγμα, το Μάρτιο φέτος η Ιταλική Πρεσβεία φετος η ελληνικη πρεσβεια εδωσε 4.000 ευρώ στο κράτος του Λιβάνου για τη βελτίωση των συνθήκων στις φυλακές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εστιαστεί σε δύο πράγματα. Υπάρχει μια μελέτη για τις βέλτιστες κατηπληκτικές για τους χώρους κράτησης και κάποια χρηματοδότηση σε συμβούλους για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί το ενδιαφέρον και η παρακολούθηση αυτής της διαδικασίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αρκεί όμως να χτίζονται καλύτερα ή μεγαλύτερα κτίρια. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που υπάρχουν για να αλλάξουν οι πρακτικές στο Λίβανο. Ο υπερπληθυσμός, 66% των υποδίκων και 30% των λαδοπών που έχουν χτίσει την ποινή έχετε ένα ποσοστό 79% κρατουμένων στο Λίβανο που δεν έχουν καταδικαστεί ή έχουν εκτίσει την ποινή τους και όμως είναι ακόμα στη φυλακή. Χρειάζονται λοιπόν καλύτερα κτίρια, αλλά πιο σημαντικό είναι να υπάρξουν πιο αποτελεσματικές διαδικασίες για να με περιορίζεται ο χρόνος κράτησης πριν από την ε, δίκη Υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις που έχουν δοκιμαστεί σε άλλα μέρη του κόσμου, η αυθαίρετη κράτηση, έχει αναγνωριστεί από, τις, από τα λιβανέζικα δικαστήρια και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό και μας προβληματίζει πάρα πολύ το θέμα των βασανιστήριων. Έχει υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο αλλά δεν έχουν προβλεφθεί ε, καθόλου εθνικές διαδικασίες εθνικές διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης. Περνάω τώρα στη Συρία. Σύντομα ο κύριος Μαλέχ θα μιλήσει πιο λεπτομερώς για μεμονωμένες περιπτώσεις. Το βασικό πρόβλημα είναι η πρόσβαση στην πληροφορία. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε πληροφορίες. Κανένας ανεξάρτητος φορέας δεν επισκέπτεται τις φυλακές της Συρία. Τα τρία προβλήματα είναι ο πολλαπλασιασμός των ε, σοφρονιστηρίων ε, και των φυλακών έχει επίσης πάρα πολλές ε, υπηρεσίες ασφαλείας. Μερικές έχουν λειτουργούν σαν χιστόρημα του Κάφκα και κάθε μία από τις υπηρεσίες αυτές έχει τους δικούς τους χώρους ε, φυλάκισης. Ορισμένοι άνθρωποι εκεί ε, βρίσκονται χωρίς να ξέρει κανένας πού ακριβώς, ε, χωρίς καμία πρόσβαση στον εξωκόσμο, επί μήνες, επί χρόνια. Δεύτερον, έχουμε πληροφορίες για πολλούς που έχουν πεθάνει ενώ βρίσκονται σε, αυτές τις, σε αυτούς τους χώρους κράτησης και πάλι δεν υπάρχει υλικό ιατροδικαστικό, δεν υπάρχουν έρευνες, οι γυναίκες συγγνώμη, και οι οικογένειε ε, είναι αναγκασμένοι πολύ γρήγορα να θάψουν τα πτώματα. Πολύ γρήγορα. Ε, μιλάμε για πολιτικούς ακτιβιστές, για bloggers, ε, ανθρώπου ανθρώπους που κρατούνται επίσης επαόριστον. Επίσης Κούρδοι και Ισλαμιστές ακτιβιστές. Το Μάιο του 2010, ε, εξετάζοντας την κατάσταση τη Συρία, υπόθηκε ότι υπάρχουν πολυάριθμες και κατ' επανάληψη περιπτώσεις ε, βασανιστήριων. Ε, δεύτερον, πολύ σύντομα, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι μία φυλακή, η Σεντνάγια, στη Συρία, που την ε, διευθύνουν οι στρατιωτικοί. Τον Ιούλιο του 2008 έγινε μια μεγάλη εξέγερση φυλακισμένων που είναι 30 χιλιόμετρα έξω από τη Δαμασκό. Είναι μια μεγάλη φυλακή. Ε, έχουμε μόνο εκτιμήσεις για τον αριθμό των ε, φυλακισμένων. υπάρχουν 2 με 3 χιλιάδες φυλακισμένοι, τουλάχιστον εκεί. Ξέρουμε ότι η εξέγερση αυτή κράτησε περίπου ένα μήνα και η σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας και περίπου 20 με 25 φυλακισμένοι σκοτώθηκαν. Γιατί μιλάω έτσι γενικόλογα. Γιατί σήμερα μετά από 2,5 χρόνια δυστυχώς δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες ε, για το τι συνέβη. Μετά από δύο χρόνια τελικά επετράπηκαν κάποιοι επισκέπτες, αλλά υπάρχει ένας κατάλογος ε, για 60 τουλάχιστον ε, κρατούμενους που δεν έχουμε καμία πληροφορία και οι Συριακές Αρχές δεν μας δίνουν καμία πληροφορεί κανένα στοιχείο για την εγκατάστασή τους. Τέλος, και θα δώσω το λόγο στον συναδελφό μου μετά από αυτό. Ε, πρέπει να μιλήσουμε για τους πολιτικούς κρατούμενους. Εκατοντάδες, οι άλλοι λένε χιλιάδες ε, ακτιβιστές, ε, πολιτικούς κρατούμενους που είναι φυλακισμένοι στη Συρία σήμερα, οι οποίοι αντιμετωπίζονται σαν ποινικοί. Συχνά παρενοχλούνται από άλλους φυλακισμένους. Δεν ξέρουμε εάν ε, εμπλέκονται και οι αρχές ή όχι, αλλά υπάρχουν πληροφορίες ότι όχι μόνο δεν έχουν επαρκή υγειονομική μέρημνα, και φυσικά οι συνθήκες κράτησής τους είναι άθλιες, αλλά ενοχλούνται και από άλλους ποινικού κρατούμενους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ εγώ για αυτές τις πληροφορίες, για την κατάσταση στο, των φυλακών στο Λίβανο και τη Συρία. Είσαστε ο βασικός ερευνητής του Human Rights Watch ε, στη Βηρητό. Και τώρα πάμε ε, κυρίως στις φυλακές στη Συρία. Θα δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή. Κυρία Πρόεδρε, Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, σα ευχαριστώ που με καλέσατε για να μιλήσω για την κατάσταση των φυλακών στη Συρία. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για αυτό το θέμα χωρί να συζητήσουμε για τι εξαφανίσει και τι ε, φυλακίσει. Ε, είναι κάτι πολύ συνηθισμένο που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70. Τώρα έχουμε πάνω από 1.700 περιπτώσει ε, από το 1979 και σήμερα. Παρότι οι εξαφανίσει αυτέ δεν, έγιναν, δεν γίνονται στην, κατά την προεδρία του Μπασάρα Παρ' όλα αυτά δεν γνωρίζουμε τίποτα ε, για τα άτομα αυτά. Από το 2000 μέχρι σήμερα ο αριθμός των φυλακισμένων γνώμης είναι περίπου 4.500. Οι περισσότεροι από, αυτού αυτούς εξαφανίζονται ε, για λίγες μέρες ή μήνες. Ε, έχουμε μερικές γνωστές περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται οπου ένα ένας χρόνο, ας πούμε απήχθη τον Οκτώβριο του, στις 14 Οκτωβρίου του 2009 ε, εξαφανίστηκε για 6 μέρε, καθώς και τη Σταλάρ Αλμαλούχη ε, χρονη blogger που ε, συνελήφθη το 2009 και δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι οι γονείς της την επισκέφτηκαν πριν από λίγες μέρες σε μια φυλακή της Δαμασκού αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό. Νιζάρα Στανάουι, μια άλλη περίπτωση, που ολοκλήρωσε μια ποινή φυλάξη πέντε χρόνια το 2009 και δεν έχει αποφυλακιστεί ακόμα. Από τότε έχει εξαφανιστεί. Ορισμένοι θεωρούν ότι δολοφονήθηκε με βασανιστήρια. Ε, ας μιλήσουμε για τα συστηματικά βασανιστήρια στις ε, φυλακές. Όταν μιλήσεις οποιονδήποτε και στους φυλακισμένους πέρα από την ε, από τη διάρκεια φυλάκιση ακούς ιστορίες για κάθε είδους βασανιστήριο. Ψυχολογικά βασανιστήρια για να αποσπαστούν πληροφορίες ε, από τις δυνάμεις ασφαλείας ε, της Συρίας. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι βασανισμού που εφαρμόζουν οι δυνάμεις ασφαλείας Παραδείγματο χάρη με νερό, με, με νερό, με τσιγάρα, με ηλεκτρικά καλώδια, ε, μαστίγωμα, ε, μαστίγωμα στα πόδια, ε, προσβολή, εκφοβισμός, εκφοβισμός και απειλές εναντίον της οικογένειας κτλ. Πολλοί Κούρδοι επίσης κρατούμενοι υφίστανται βασανιστήρια. Ορισμένοι πέθαναν με βασανιστήρια. Δεν έχουμε πλήρη κατάλογο και δεν μπορώ να σας τα πω λόγω έλλειψης χρόνου. Μάμο Κάνζο ε, ήταν ένα άτομο το οποίο στις 15 Μαρτίου του 2008, 4 ε, συγγνώμη, ε, κρατήθηκε, χτυπήθηκε με ένα φοβερό όπλο στο κεφάλι και άνοιξε το κεφάλι του με μία πληγή χένουσα 10 εκατοστών αυτές ε, πήγε στο νοσοκομείο, αλλά εκεί είδαν οι γιατροί ότι είχε πάρα πολλά σημάδια από συστηματικό βασανισμό. Επίσης, ε, παραπονέθηκε για πόνους στο κεφάλι, για αίσθηση έλλειψης ισορροπίας και το Μάιο ε, του 2004 πέθανε λόγω εσωτερικής ομορραγίας στον εγκέφαλο που προκλήθηκε από συστηματικό συστηματικά χτυπήματα λόγω της αυθαίρετης αυτής κράτησης. Ο Φεράς Μαχμούτ Αμπταλάχ σκοτώθηκε στη στρατιωτική φυλακή της Δαμασκού όπου ήταν υπό ανάκριση τον, ε, τον Ιανουάριο 2000, από το 2004. Τον Ιανουάριο 2009 δώσαν το σωρό του στην οικογένειά του τέσσερις μήνες μετά από την αυθαίρετη κράτησή του με την υποψία και μόνο ότι ήταν Ισλαμιστής το απόγευμα της ίδιας μέρας είχε ταφεί, η οικογένεια του δεν μπόρεσε να κάνει μια πραγματική διαδικασία τα... ταφής και επρόκειτο για ένα άτομο το οποίο είχε γεννηθεί το 1966. Ένα, μια άλλη περίπτωση, ένας ε, πατέρας τεσσάρων παιδιών εξαφανίστηκε το 2007 σε μια περιοχή της ε, Δαμασκού που είναι γνωστή ως Ρουχνέτη. Το σταμάτησε η ασφάλεια, η κρατική ασφάλεια, μπροστά στη γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά του βγάλαν από το αυτοκίνητό του και τον δίραν μέχρι θανάτου στον δρόμο. Μια άλλη περίπτωση, ένα άτομο 33 χρονών, παντρεμένο και πατέρα ενό παιδιού, ο οποίο εργαζόταν στη Δαμασκό, κρατήθηκε για 40 μέρε ε, κατηγορούμενος για κλοπή χρημάτων από την τράπεζα που εργαζόταν και βασανίστηκε εν κρατήσει κάτι που δείξε στο θάνατό του το 2008. Η ισορός του δόθηκε στην οικογένειά του δύο μέρες αργότερα. Ο Σιλάλ Χαουράν Αλπαβέση στην Δαμασκό το 1971 γεννήθηκε και σκοτώθηκε στις 31 Μαΐου του 2010 ενώ τελούσε υπό παράνομη κράτηση στην φυλακή ασφαλείας της Δαμασκού και υπέστη κακομεταχείριση πριν από το θάνατό του. και μου είπανε τα εξής από ένα ο οποίος ε, πέρασε σε, εξαφάνιση ότι τον βασανίσανε με λοστούς και άκουσα τις κραυγές τους με τα ίδια μου τα αυτιά και χρησιμοποιήθηκαν επίση ηλεκτρικά καλώδια τα οποία χρησιμοποιούντο και ένας, ε, ένα μεταλλικό κουτί το οποίο είχε Είχε φωτιά μέσα, δεν ξέρω πώς χρησιμοποιούνται όλα αυτά, μου είπε. Οι καταστάσεις κράτησης είναι αποτρόπες. Είναι σε 60 τετραγωνικά μέτρα 60 άτομα. Για να μπορέσει κανείς να πάει στην τουαλέτα πρέπει να περάσει πάνω από τους άλλους κρατουμένους και να τους πατήσει. Δεν έχει τη δυνατότητα ένας κρατούμενος εκεί να είναι σε επαφή με τους ε, δικηγόρους του και ορισμένοι κρατούμενοι πάντα βρίσκονται συνοδευόμενοι από κάποιον ε, φρουρό της φυλακής. Δεν έχουν το δικαίωμα να πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη της ε, φυλακής και δεν μπορούν να έχουν έγγραφα ή βιβλία μαζί τους. Είναι φυσικά διαφορετική η κατάστασή τους και το γράμμα που έχετε πάρει από τη φυλακή της Άκρα <clears throat> περιλαμβάνει ε, και άλλες περιπτώσεις όπως έχει αναφέρει η Amnesty International. Είναι πάρα πολλές αυτές τις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται σχεδόν σε κάθε τετράγωνο ένα υπόγειο για κράτηση και βασανιστήρια. Δεν πρόκειται να σας αναφέρω όλο το κατάλογο επειδή δεν έχουμε χρόνο. Είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος, πολύ μακρύς ο κατάλογος των κέντρων κράτηση στη Συρία. Πριν κλείσω όμως, θέλω να αναφέρω ότι είναι πολύ δύσκολος αγώνας των ε, δικηγόρων που προσπαθούν να υπερασπιστούν τους ε, κρατουμένους. Υπάρχει απόλυτη ατιμορρησία για αυτούς οι οποίοι κάνουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι δικηγόροι παρενοχλούνται από τις ε, αστυνομικές αρχές και επίσης και από το δικηγορικό σύλλογο, ο οποίος δεν είναι ανεξάρτητος, αλλά είναι βραχίωνας του καθεστώτος. Ε, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, ένας ε, δικηγόρος, επειδή παρακολούθησε τις διαδικασίες σε κάποιο δικαστήριο, κρατικό και επειδή πληροφόρησε μια, υπο, μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του αφαίρεσαν το δικαίωμα άσκησης της δικηγορία διαβίου. Επίσης, πολλές φορές δεν υπάρχει, δεν δίνεται άδεια στους δικηγόρους να επισκεφθούν του πελάτες τους για να συζητήσουν τις περιπτώσει αυτές. Εγώ ήλπιζα ότι μετά από το θάνατο χαφέ Αλασάτ είχε αλλάξει προ το καλύτερο κατάσταση στη Συρία. Αλλά όπω έχετε ακούσει και εσείς και εγώ από αυτούς που είναι στη Συρία, η κατάσταση παραμένει όσο αποτρόπια ήταν στο παρελθόν και επιδεινώνεται ακόμα. Μου είπαν ορισμένοι ότι η κοινωνία της Συρίας είναι έτοιμη να καταρρεύσει. Σα συγκετεύω να κάνετε ό,τι είναι δυνατό και βάσει τη συνείδησή σας να βοηθήσετε το λαό τη Συρίας να αποκτήσει τα ελάχιστα δικαιώματα τα οποία πρέπει να έχει. Ο λαός της Συρίας είναι ο φίλος που χρειάζεστε και όχι η κυβέρνηση της Συρίας. Αύριο συζητάει η Κομισιόν με εκπροσώπους της Συρίας για την συμφωνία σύνδεσης με τη Συρία. Το να γίνει τώρα μια συμφωνία με ένα ε, εγκληματικό καθεστώς θα κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση συνένοχο σε αυτά τα εγκλήματα. Είναι σημαντική η συνεργασία με τη Συρία, αλλά όχι σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει. Ευχαριστώ. Μας δώσατε εντυπωσιακέ λεπτομέρειες για τις μεθόδους βασανισμού στις ε, φυλακές ε, και σοφονιστήρια της Συρίας. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ακούσουμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να σταματήσει αυτή η ολέθρια πρακτική και η κακομεταχείριση, τα βασανιστήρια των φυλακισμένων στο Λίβανο και τη Συρία. Φυσικά, θέλω να πω σε όλους ότι και άλλες χώρες χρησιμοποιούν αυτές τις απάνθρωπες μεθόδους, αλλά σήμερα η προσοχή μας στρέφεται στο Λίβανο και τη Συρία. Αργότερα θα μιλήσουμε και για την κατάσταση των φυλακών στο Ισραήλ και στο, στην Παλαιστίνη. Ε, σας εξήγησα στην αρχή ότι δεν μπορέσαμε να σήμερα να καλύψουμε αυτό το θέμα γιατί δεν είχαμε τους ομιλητές. Ε, δίνω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας πει την άποψή της και να σχολιάσει αν μπορεί για τη συμφωνία που μας ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής. Τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, που οργανώνετε αυτή την ακρόαση. Ευχαριστώ τους δύο ομιλητές που μας έδωσαν τόσα πολλά στοιχεία συμφωνούμε και συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που αναφέρατε. Ε, Ιδίω ε, ας ξεκινήσουμε με τη Συρία για του ε, τους ισχυρισμούς για κακομεταχείριση, ε, την εξαφάνιση, τις τους βασανισμούς, τις κακές συνθήκες κράτησης, έλλειψη βασμού προς τους κρατούμενους κτλ. Αυτό δείχνει ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία δεν έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και δείχνει ότι υπάρχουν σοβαρότατες ανακρίβειες ε, και έλλειψη συμμόρφωσης της Συρίας με τις δεσμεύσεις της ε, με βάση το, τη σύμβαση κατά του βασανισμού και το, τη συμφωνία του ΟΗΕ για τα, ανθρώπιν, για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα. Έχουμε πάρα πολλούς κρατούμενους, ε, ε, συνείδησης, ε, απόψεων όπως ε, bloggers, δικηγόρους, ακτιβιστές κτλ. Η Συρία έχει γίνει μια δήλωση μάλιστα, μια έκκληση προς τη Συρία για να σεβαστεί τα, τις δεσμεύσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Την περασμένη εβδομάδα, στις 18 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του επικεφαλής του γραφείου της στη Συρία επανέλαβε διάφορες δηλώσεις δημόσια ε, καθώς ο κύριος Χαλ Χασάν ε, πήρε ένα πολύ διακεκριμένο βραβείο. Φυσικά είμαι απογοητευμένος για την ε, αρνητική απόφαση του εφετείου ε, της υπόθεσης του κυρίου Χαλ Μασάλ. Εμείς ε, θα μιλάμε για την περίπτωση αυτού και για άλλες περιπτώσεις όπου η Συρία δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα επανερχόμαστε σε αυτό το θέμα, σε όλες τις επαφές μας με τη Συρία και η αντιπροσωπεία μας ε, εκεί και η πρεσβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τεμασκό παρακολουθεί την κατάσταση, τις δίκες και προσπαθεί να μιλήσει για τις καλές πρακτικές για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το χρηματοδοτικό μέσο για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία δίνει ε, βοήθεια για τη μεταρρύθμιση της ε, δικαιοσύνης και για τον ενθαμωμένο διάλογο με την... Ε, αυτό έγινε για τη δικαιοσύνη πέρυσι και φέτος για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και την ε, κυβέρνηση. Ε, από το 2009 ε, δεν έχουμε υπογράψει αυτή τη Συμφωνία εταιρική Σχέσης και Συνεργασίας γιατί αξιολογούμε τις πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις της συμφωνίας αυτής. Θέλω να επαναλάβω ότι με βάση την εμπειρία που έχουμε από την πολιτική γειτονία στην περιοχή, θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία συνεργασίας είναι ένα μέσο για να θεσπίσουμε ένα σταθερό πολιτικό διάλογο με τη Συρία ε, και κυρίως για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις ε, στην περιοχή ε, διαπιστώσαμε ότι με αυτόν τον τρόπο βάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ατζέντα ούτως ώστε να συζητούμε με τις χώρες. Τώρα, για το Λίβανο. Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κομβικό σημείο στις σχέσεις μας. Υπάρχει ένα σχέδιο δράσης ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Λιβάνου για, όπου υπάρχουν και δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα για μια ανεξάρτητη και ελεύθερη δικαιοσύνη και εφαρμογή των αποφάσεων της δικαιοσύνης, καταπολέμηση του βασανισμού και εστίαση στην εφαρμογή της συμφωνίας του ΟΗΕ. Έχουμε λοιπόν συμφωνημένο αυτό το σχέδιο δράση. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτω ώστε να έχουμε τακτικό διάλογο με το Λίβανο. Ούτω ώστε να δούμε τι πρόοδος έχει σημειωθεί σε αυτή τη χώρα. Τελευταία φορά ε, συνεδριάσαμε την Επιτροπή, τη σχετική αυτή επιτροπή το Μάιο στη Βηρητό και πάντα συζητάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα με το Λίβανο. Εκεί ακούμε περιπτώσεις βασανισμού, ε, κακομεταχείρισης. Ε, συζητήσαμε την έλλειψη συμμόρφωσης ε, του ποινικού κώδικα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση κατά του βασανισμού, την οποία έχει προσυπογράψει η Συρία. Η, Συμβία, η Συρία και η πρόσβασή της στο προαιρετικό πρωτόκολλο κατά του βασανισμού που υπογράφηκε το 2008 ήταν ένα θετικό βήμα όμως ο Λίβανος ακόμα δεν έχει τους μηχανισμούς πρόληψης όπως ε, προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Παρακολουθούμε την κατάσταση. Ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε είναι ε, η σύμβαση κατά του βασανισμού που ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές ε, και το πώς το εφαρμόζει ο Λίβανος. Ένα άλλο θέμα είναι η μονάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, η οποία είναι υποεπανδρομένη λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα. Επίσης η μεταφορά του, της ευθύνης για τις φυλακές προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ελπίζουμε ότι αυτή η κίνηση θα βελτιώσει την κατάσταση στις φυλακές, αλλά φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν και επαρκείς πόροι για να είναι θετικό αυτό το βήμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπίστωσε ότι υπάρχουν θετικά βήματα στο Λίβανο. Όταν ο Επίτροπος ε, επισκέφθηκε αυτή τη βδομάδα το Λίβανο, ε, εκινήσαμε δύο, ε, μια διαδικασία χορήγησης 2 εκατομμυρίων ευρώ ε, για τον εκμοντερνισμό των, ε, του σοφρονιστικού συστήματος. Επίσης για την υποστήριξη μη κυβερνητικών οργανώσεων που υποστηρίζουν και βοηθούν τις οικογένειες αλλά και τα θύματα εξαφανίσεων και κρατήσεων. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλέσω την κυρία να πάρει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους προσκαλεσμένους μας οι οποίοι μας έδωσαν πολλές πληροφορίες για το Λίβανο την επόμενη εβδομάδα θα συμμετέχω σε μια επίσημη αντιπροσωπεία την αντιπροσωπεία του Μασρέκ που θα μεταβεί για μια ολόκληρη εβδομάδα στο Λίβανο. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Βηρητό. Θα επισκεφθούμε ένα καταβλισμό Παλαιστινίων προσφύγων δεν θα επισκεφθούμε φυλακές, αλλά πιστεύω ότι τα στοιχεία που ακούσαμε ήταν πολύ σημαντικά διότι έχουμε προβλέψει συναντήσεις, επαφές με τον Υπουργό Εσωτερικών Δικαιοσύνης και Άμυνας και δεσμεύομαι ως μέλος της Υποεπιτροπής ότι θα συζητήσω για την κατάσταση στις φυλακές του Λιβάνου με τους εκπρόσωπους της κυβέρνησης στη διάρκεια αυτής της επίσκεψης αντιπροσωπείας μα. Μία ερώτηση για τον κύριο Ουρή. Θα μπορούσε να μας δώσει λίγα περισσότερα στοιχεία για τους αλλοδαπούς που κρατούνται στις φυλακές που αποτελούν ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό του, των τροφίμων. Μπορεί να μας αναλύσει τις χώρες προέλευσης αυτών των αλλοδαπών κρατουμένων. και ποια είναι τα εγκλήματα ή τα δικήματα τα οποία έχουν αυτή διαπράξει. Τώρα, για τη Συρία. Αναφέρθηκε η κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων και ο αριθμός τους. Η Human Rights Watch αναφέρει ότι υπάρχει καμιά εκατοστή πολιτικών κρατουμένων, αλλά αναφέρονται και χιλιάδες άτομα, τα οποία υπο... φαίνεται ότι κρατούνται διότι είχαν κάποιες σχέσεις με κουρδικές οργανώσεις ή ανήκουν σε οργανώσεις αντιπολίτευσης ή της κοινωνίας των πολιτών. Πολλοί βρίσκονται στη φυλακή βρίσκονται στις ε, φυλακές των υπηρεσιών ασφαλείας, οι πολιτικοί κρατούμενοι. Ε, ε, δικάζονται από ειδικά, δικαστήρια χωρίς να έχουν δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Έχετε να μας δώσετε πληρωματικές πληροφορίες για αυτά τα θέματα. Διότι η περίπτωση για την περίπτωση του κυρίου Αλμάλεχ. Η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και ότι αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται όλες τις ευκαιρίες που της παρέχονται για να αναφέρεται σε αυτή την περίπτωση αλλά και σε άλλες. Ο κύριος Μάλεχ είναι στη φυλακή εδώ και ένα χρόνο και ακούμε τις ίδιες δηλώσεις στις απαντήσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα χωρίς να αλλάζει τίποτε. Όλα αυτά τα διαβήματα λοιπόν, όλες αυτές οι προσπάθειες από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Τα κράτη-μέλη και η ύπατη ε, εκπρόσωπος θα μπορούσαν ενδεχομένω να σκεφτούν άλλα μέτρα και απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιε είναι οι άλλε δράσει που θα μπορούσαν να αναλάβουν η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ώστε να καταλήξουμε σε ένα πιο θετικό αποτέλεσμα. Θα, θα μπορούσατε να συναντηθείτε στη Βηρητό, διότι ο κύριος Γούρι έχει, την έδρα του στη Βηρητό και θα μπορούσατε να τον συναντήσετε εκεί και να σας δώσει όλα τα στοιχεία που θέλατε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος είναι ο ακριβής τίτλος. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Είμαι πολύ ευτυχής που αποφασίσατε να οργανώσετε αυτή την ακρόαση. ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεδομένου ότι ο εκπρόσωπος μας είπε ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Συρία. Και όμως η Επιτροπή εφαρμόζει, ετοιμάζεται να υπογράψει μια συμφωνία ε, γειτονίας. Με εκπλήσει αυτό. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο μετά από όλες τις λεπτομέρειες που ακούσαμε σήμερα το πρωί, σήμερα το απόγευμα εδώ, για τον τρόπο, για τη συμπεριφορά ε, ε προς τους φυλακι... για το, τη μεταχείριση των φυλακισμένων, την εξαφάνιση μερικών κρατουμένων. Πώς είναι δυνατόν να υλοποιηθεί ένας αποτελεσματικός διάλογος που θα περιλαμβάνει, που θα περιλαμβάνει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ποιο σημείο η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει προσπαθήσαμε να κάνουμε ανοίγματα, προσπαθήσαμε να διευρύνουμε τις σχέσεις μας προσφέροντας εμπορικές ε, ε, διευκολύνσεις λοιπά, Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν έφερε αποτελέσματα, οπότε θα πάψει πλέον να ισχύει η συμφωνία. Πότε επιτέλους θα πείτε όχι και θα θέσετε ένα τέρμα σε αυτή τη συμφωνία, εφόσον δεν φέρνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Ντερόσα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ουριέν, τον κύριο Ελ Μάλεκ και μετά στην αλλά έχουμε άλλη μια χώρα που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Για το θέμα των ξένων, ο αριθμός των μη Λιβανέζων που είναι στη φυλακή είναι περίπου 35%. Είναι πολλοί ξένοι οι οποίοι εκτείουν την ποινή τους. Από τα 35% 16% είναι Παλαιστίνοι και Σύριοι. Είναι εγκατεστημένοι στο Λίβανο για πολύ καιρό. Αλλά τα υπόλοιπα 19% είναι από διάφορες εθνικότητες, η μεγαλύτερη ομάδα είναι, με μεγαλύτερες ομάδες είναι από το Σουδάν, πολίτες του Σουδάν και μεταξύ των γυναικών είναι οικιακές βοηθοί που έρχονται από τις Φιλιππίνες, Λάνκα, Αιθιοπία, Νεπάλ. Γιατί είναι στη φυλακή τώρα. Ο κύριος λόγος για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους είναι επειδή δεν έχουν ε, έγγραφα, νόμιμα έγγραφα διαμονής. Πολλές φορές δεν φταίνε γιατί οι εργοδότες τους τους παίρνουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και τα έγγραφα διαμονής. Αλλά ο δεύτερος λόγος είναι μικροαγκλήματα, μικροαδικήματα όπως κλοπές κτλ. Θα μπορούσα να σας δώσω και περισσότερες λεπτομέρειες για όλα αυτά, αν θέλετε. Για τα έκτακτα δικαστήρια στη Συρία. Πράγματι, υπάρχει το ανώτατο δικαστήριο κρατικής ασφάλειας, το οποίο δημιουργήθηκε βάσει ενός νόμου εκτάκτης ανάγκης. Από ό,τι ξέρουμε, καταδικάζει τουλάχιστον 250 άτομα κάθε χρόνο. Μπορεί να υπάρχει και ένα δεύτερο τέτοιο δικαστήριο το οποίο θα ξεκινήσει βάσει των πληροφοριών που έχουμε. Είναι προφανώς ένα δικαστήριο το οποίο δεν σέβεται καμία διαδικασία. Υπάρχει ένας δικαστής σε αυτό το δικαστήριο, ο οποίος έπρεπε να είχε συνταξιοδοτηθεί πριν από 8 χρόνια, αλλά είναι ακόμα εκεί. Οι περισσότεροι Κουρδιστές, Κουρ, Κούρδοι ακτιβιστές, συγγνώμη, θεωρούνται ύποπτοι για Ισλαμιστική δράση, αλλά και πολιτικοί ακτιβιστές και άνθρωποι με ιστολόγια έχουν καταδικαστεί από αυτό το δικαστήριο και δεν είναι απλώς ότι δεν βελτιώνεται η κατάσταση. Δεν βλέπουμε να υπάρχει παραμικρή βελτίωση στην πρακτική αυτού του δικαστηρίου και είναι ένα από τα κύρια προβλήματα στη Συρία. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν, κλείνοντας, το πραγματικό ερώτημα είναι ποια είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική εναντί της Συρίας. Αυτό είναι το ουσιαστικό, το κέριο ερώτημα εδώ. Γιατί υπήρξαν πολλές δηλώσει ότι όλοι είναι, με... όλοι είναι απογοητευμένοι ότι δεν μπορούν να ασκήσουν πίεση πάνω στη Συρία αλλά εδώ νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο αμφισβητώντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητώντας να υπάρξουν συγκεκριμένα βήματα. Ξέρουμε ότι η στρατηγική που ακολουθεί μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει λειτουργήσει. Είναι καιρός να σκεφτούμε εναλλακτικέ στρατηγικές. Ο κ. Αλμάδε. Σας ευχαριστώ. Δύο ερωτήματα που μπορώ ίσως να σχολιάσω. Καταρχήν ο αριθμός των κρατουμένων τα στοιχεία που έχω εγώ και εδώ συμφωνούν σχεδόν όλοι οι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα και έξω από τη Σύρια 4.500 ε, κρατούμενοι συνείδησης και 17.000 άτομα τα οποία έχουν εξαφανιστεί σε διάφορες χρονικές στιγμές. Για τις δικαστικές τώρα διαδικασίες. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να σας δώσει μια σαφή εικόνα για το πώς γίνεται <clears throat> αυτή η διαδικασία. Γιατί κοιτάζοντας δύο παρόμοιες περιπτώσεις του πατέρα μου και ενός άλλου, που ήταν και οι δύο δικηγόροι με αντιμετωπίζοντας την ίδια κατηγορία, την διασπορά ψευδών ειδήσεων, στην περίπτωσή τους ο ένας, ο πατέρας μου, δικάστηκε σε στατηγικό δικαστήριο, ο άλλος σε ένα πολιτικό δικαστήριο. Πήρανε και οι δύο την ίδια ποινή. Τρία χρόνια φυλακή. Γιατί γίνεται αυτό με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ποτέ δεν βρέθηκε στο στρατό στη ζωή του. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε 10 χρόνια που φέρεται ενώπιον στρατι... στρατιωτικού δικαστηρίου 2000-2004-2010. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς επιλέγουν ποιους κατουμένους θα δικάσουν σε ποιο δικαστήριο. Αλλά τελικά οι ίδιες ποινές απαγγέλλονται εναντίον τους είναι έτοιμες οι ποινές αυτές. Ξέραμε ποια ήταν η ποινή για τον Μοχάμετ Αλχάσανη, προτού τον καταδικάσαμε, ξέραμε την επόμενη μέρα ότι θα τον καταδικάζαν σε τρίτη φυλάξη. Αυτό συμβαίνει συνέχεια. Σας ευχαριστώ κύριε Χέρτς. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο βουλευτές για τα ερωτήματά τους, τα οποία είναι απόλυτα λογικά και φυσικά είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο ερωτήματα. Είναι το θέμα του πώς μπορούμε να ασκήσουμε πίεση, πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επαφή σε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο με την κυρία Άστον και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα από τα ψηφίσματά του ζητά να έχει πρόοδο στη Συρία και τα αποτελέσματα είναι μέχρι στιγμής πάρα πολύ συχνά. Η συζήτηση για τη Συμφωνία Σύνδεση με τη Συρία χρονίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι μια συζήτηση ανάλογη με το δίλημα της κότας ή του αυγού. Πρέπει να μην έχουμε συμφωνία σύνδεσης λόγω της έλλειψης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή η απουσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία που θα μας δώσει εργαλεία να δράσουμε. Υπάρχουν λοιπόν απόψεις και υπέρ και κατά, το γνωρίζω αυτό Απλώς <clears throat> εγώ θα σας παραθέσω αυτά που λέει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου. Στο σημείο 7 λέει το Κοινοβούλιο ότι βλέπει την προοπτική μια συμφωνία σύνδεσης ότι θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για να αντιμετωπιστούν και τα θέματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμών και την ενίσχυση τη διαδικασία μεταρρύθμιση στη Συρία και επομένω καλεί την Κομισιόν και το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει αυτό τον κέριο μοχλό για να υπάρξει μέσω ενό σχεδίου δράσης για την ε, δημοκρατία που καθορίζει τελείω και πλήρω τι προόδου που θέλει να επιτύχει από την πλευρά της Συρίας. Αυτό με πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Βέβαια, ο δρόμος από την υπογραφή μιας συμφωνίας ω την κύρωσή τη από τα κάτι μέρη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι, μπορεί να είναι μάλλον, πολύ μακρός χρόνος και αυτό είναι χρόνο ο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όπως ε, ακούσαμε σήμερα υπάρχουν πραγματικά πάρα πολύ αξιόπιστες ιστορίες αυτοπτών μαρτύρων για την κατάσταση εκεί και επομένω έχουμε κάθε λόγο να θίξουμε τα θέματα αυτά και πάλι στο μέλλον. Και να μην ξεχάσουμε το Λιβάνο και τη Συρία. Λοιπόν, Ευχαριστώ και πάλι, σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε. Δεν θα εγκαταλείψουμε τελείως το θέμα. Από το Διεθνές Σύμφωνο Πολιτικών και Αστικών Δικαιωμάτων όλοι όσοι στερούνται ελευθερίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με ανθρωπισμό και σεβασμό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα ήθελα να το πω αυτό διότι ο συνάδελφος Χίγκης είναι εδώ και θυμάστε ότι πριν από λίγες εβδομάδες ήταν εδώ και δια, έχοντας διαπιστώσει σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε μια χώρα, σε μια χώρα που ασκεί αυτή τη στιγμή την προεδρία του ΟΑΣΕ, το Καζακστάν. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα στο θέμα στο επόμενο θέμα που είναι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν. Στην αρχή της συνεδρίασής μας για όσους δεν ήταν παρόντες θύμισα ότι η ακρόαση δεν αναβλήθηκε λόγω της επίσκεψης του Προέδρου Καζακστάν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά μετά από αίτηση του Προέδρου του Κοινοβουλίου μεταφέρθηκε από την Τρίτη στη Δευτέρα, διότι αύριο ο Πρόεδρος Μπούζεκ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του, Αζερ... του Καζακστάν. Θα ήθελα να αναφέρω ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου πρόσφατα ψήφισε ένα ψήφισμα, μια πρόταση ψηφίσματος για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΑΣΕ, καλώντας το Καζακστάν πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσει ε, την προστασία ορισμένων σημαντικών αξιών, ελευθερία έκφρασης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, φαντάζομαι ότι εκφράζω τα αισθήματα όλων μας λέγοντας ότι αυτά θα χρειαστεί να γίνουν γρήγορα. Το Καζακστάν προωθεί την υποψηφιότητά του για μια θέση στη Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την περίοδο 2012-2015. Και θα ήθελα να προσθέσω συνάδελφοι ότι από τον συνάδελφο Στίβενσον, τον ειδικό εκπρόσωπο του, της Προεδρίας του ΑΣΕ για τα οικολογικά και περιβαλλοντικά θέματα, έλαβα μία επιστολή, την οποία υποσχέθηκα ότι θα σας ε, αναφέρω εν συντομία. Λέει στην επιστολή του ότι το Καζακστάν υπογράμμισε την πρόληψη συγκρούσεων, την κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος και τις διεθνείς μεταφορές σαν σημαντικά θέματα. Θα φιλοξενήσουν μία σύνοδο κορυφή στην Αστάνα του ΟΑΣΕ το Δεκέμβριο, στην οποία 56 κράτη-μέλη θα συμμετέχουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Θα είναι η πρώτη φορά που μία σύνοδος κορυφής, έχει γίνει μία σύνοδο κορυφή του ΟΑΣΕ. Νομίζω από το 1999 έχει να γίνει άλλη τέτοια σύνοδο κορυφή. Ο συνάδελφος Στίβενσον προσθέτει ότι το Καζακστάν η πιο ανεπτυγμένη οικονομία των πέντε ε, δημοκρατών της Κεντρικής Ασία, έχει ανοίξει την οικονομία της στις επενδύσεις και είναι εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον ως χώρα. Τώρα, περνάμε στην ακρόαση. Ε, Έχουμε την κυρία Ζακλίν Χέιλ, η Χάρλ, δεν ξέρω πώς προφέρεται το όνομά της. Η κυρία Ζέκλιν Χιούμ από το Ινστιτούτο Ανοιχτή Κοινωνίας, που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κεντρική Ασία, η οποία θα μας μιλήσει και την κυρία Αντριάννα ε, Μπέργα από τη Human Rights Watch και είμαστε επίσης ιδιαίτερα ευτυχείς που έχει, ε, μία μη από το Καζακστάν που ήταν προσκεκλημένη μπόρεσε, μπόρεσε να έρθει παρόλε τις δυσκολίες και ο εκπρόσωπός της θα πάρει επίσης το λόγο. So, uh, uh, uh, Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον δόκτορα So Με το πρόσωπο της Human Rights Watch. Το κείμενό σας θα το μοιράσουμε, αλλά προτιμάμε να μας μιλήσετε ελεύθερα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ που τη Human Rights Watch σε αυτή την ακρόαση. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση του Καζακστάν έλαβε θετικά σημαντικά μέτρα επικύρωσε τη, τα μέσα προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και εφαρμόζοντα κάποιε μεταρρυθμίσει στο σύστημα ποινική δικαιοσύνη. Αλλά στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά δεν έχουν συμβεί στην πράξη ουσιαστικέ μεταβουλέ. Στη διάρκεια τη προεδρία του, του ΟΑΣΕ του 2010, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχει στασιμότητα στο Καζακστάν ή και οπισθοδρόμηση έχουν περιοριστεί ε, οι περιορισμοί που επιβάλλει η νομοθεσία για την ελευθερία των μέσων ενημέρωση εξακολουθούν να ισχύουν. Τιμωρεί τους ακτιβιστές η κυβέρνηση ε, επειδή παραβιάζουν ορισμένες ε, απαγορεύσεις. Το 2010 ο Ευγένη Ζόφτετ, ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σημαντικότερο ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Καζακστάν, είναι ακόμα στη φυλακή. Οι δημοσιογράφοι που επικρίνουν τι πρακτικέ και την πολιτική τη κυβέρνηση υφίστανται απειλέ, ε, ε, διάφορε κυρώσει ε, αστικέ. ή ποινικέ. Σύμφωνα με το, έναν οργανισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Καζακστάν το 2010. Πέντε δημοσιογράφοι δέχθηκαν σωματική επίθεση και άλλοι πέντε κατηγορήθηκαν για ποινική δυσφήμιση. Την 1η Μαρτίου του 2010 ο επικεφαλής της κρατική υπηρεσίας για την, την επικοινωνία και τα δίκτυα δήλωσε ότι υπήρχε, υπήρχε ε, ε, ε, είχε προκύψει ένα πρόβλημα στα ηλεκτρονικά συστήματα. Επίσης, οι θρησκευτικές, ε, τα οι ιστοσελίδες ε, κατά πάσα πιθανότητα επίσης, επίσης πρόκειτο να καταργηθούν. Επίσης, η σελίδα της ανεξάρτητης εφημερίδας Ρεπούμπλικα. Τον Ιούλιο του 2010 οι αρχές αρνήθηκαν στον Ραμαζάν Γκερμπεγιόφ, εκδότη της εφημερίδας Αλταφόρ, να, να τον ελευθερώσουν παρόλο που είχε κτίσει μέρος της ποινή του. Η ποινή του ήταν τρία χρόνια, το 2009, επειδή είχε αποκαλύψει δήθεν μυστικά κρατικά, διότι είχε δημοσιεύσει η εφημερίδα του μία επιστολή στην οποία η υπηρεσία εμφανιζόταν να προσπαθεί να πείσει ε, να αλλάξει την απόφασή του ένα δικαστήριο. Η δίκη δεν ήταν ανοιχτή στο κοινό και δεν είχε πρόσβαση σε δικηγόρο της επιλογής του. Σε ό,τι αφορά την ελευθερία του συνέρχεστε, το Μάρτιο του 2006 ο Βλαντιμίρ Κοσλόφ, ο ε, σημαντικότερος ακτιβιστής του κόμματος ΑΛΚΑ, συνελήφθη Οι κατηγορίε του απαγγέλθηκαν επειδή είχε μοιράσει φυλάδια που επέκριναν τη δίκη του Μουχτάρ Τακίτσεφ, πρώην διευθυντή τη κρατικής πυρηνικής εταιρείας, του οποίου η φυλάκιση πολλοί πίστευαν ότι οφείλεται σε πολιτικά κίνητρα. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον, το Κοσλόφ είχε μοιράσει τα φυλάδια σε, μια, σε ένα πεζόδρομο στο Αλμάτι. Άλλοι που κάναν το ίδιο με εμπορικά φυλάδια την ίδια στιγμή δεν συνελήφθησαν. Στις 2 Μαΐου 2010 ο Γερμέγ Ναρεμπάγεφ, επικεφαλής του κοινωνικού ε, κινήματος Dream, ε, καταδικάστηκε σε σύλληψη διότι είχε συμβάλει στη συγκέντρωση 500 ατόμων. Μετά τη σύλληψή του κατηγορήθηκε ε, ότι αντιστάθηκε στην αστυνομία. Στις 23 Ιουνίου το δικαστήριο τον καταδίκασε σε τετραετή φυλάκιση. Τον Ιούνιο τα δικαστήρια τιμώρησαν πέντε άτομα, ακτιβιστές και δημοσιογράφους, ότι δήθεν είχαν οργανώσει και είχαν λάβει μέρος σε μη επιτρεπόμενες ε, συνεδριάσεις και συναντήσεις. Τα άτομα, τα αυτά είχαν οργανώσει μια πολύ μικρή διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία του Αλμάτι για το γεγονός ότι είχε ε, διαβίου, ε, διαβίου ασυλία στον πρόεδρο. Το 2010 γιορτάστηκε ολοκληρώθηκε το πρώτο έτος της φυλάκισης του Ζόφτες, ο οποίος το 2009 διευθυντής του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κράτους Δικαίου του Καζακστάν θεωρήθηκε ύποπτος για ανθρωποκτονία μετά από μια δίκη δίκη. Καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια σε μια φυλακή αγροτική που του εξασφάλιζε κάποια ελευθερία κινήσεων. Εκείνος επέλεξε να μην κάνει χρήση αυτής της, ε, αυτής της ελευθερίας. Η Human Rights Watch έχει δημοσιεύσει επίσης εκθέσεις για τη μεταχείριση των αγροτών στο Καζακστάν. δεν τους δίνουν, οι εργάτες αυτοί εργάζονται ε, για τη συλλογή καπνού για λογαριασμό της εταιρείας Philip Morris. Αυτοί οι εγρότες υποχρεώνονται σε πολλές περιπτώσεις να κάνουν καταναγκαστική υποχρεωτική εργασία, δεν ε, τους αφαιρούνται τα χαρτιά τους και επίσης μεταξύ αυτών είναι και παιδιά. Υπάρχουν πολλοί φοβερές περιπτώσεις εκμετάλλευσης, εκμετάλλευσης παιδιών τα οποία υποχρεώνται να εργαστούν σε πολύ μικρή ηλικία και κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Η Φίλιπ Μόρις έχει υπογράψει συμβάσεις με τους γεωργούς εξασφαλίζοντας, θέλοντας να εξασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι εργάζονται πλέον κάτω από κανονικές συνθήκες. Έχουν εφαρμόσει επίσης ένα σύστημα υποβολής παραπώνων για τους υπαλλήλους και τους αγρότες που εργάζονται για τη Φίλιπ Μόρις στο Καζακστάν και προσπαθεί να συνεργαστεί, να συνεργαστεί με την ώστε να υπάρχει ε, δυνατότητα πρόσβαση σε σχολική εκπαίδευση στα παιδιά των αγροτών και να αποφεύγεται η υποχρεωτική εργασία για τα παιδιά. Ένα συνασπισμός από από το Καζακστάν και άλλων χωρών είχε σκοπό να οργανώσει μια συνδιάσκεψη στην Αστάνα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΑΣΕ. Η παράλληλη διάσκεψη έχει σκοπό να αποτελέσει μια πλατφόρμα για τις ομάδες της κοινωνίας ε, των πολιτών για την χάραξη στρατηγικής που θα ενισχύσει τον ΟΑΣΕ για τους μηχανισμούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα περιλαμβάνεται στην επίσημη ατζέντα, αλλά θα υπαρέχει μια δυνατότητα, θα παρέχει τη δυνατότητα σε όλους ε, θέλουν να εκφραστούν για τον τρόπο με τον οποίο θα, μπορούσε να θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει ο ΑΣΕ. Ζητήθηκε τον Γιούριο Μπλάτσα από την κυβέρνηση να καταργήσει ε, να ακυρώσει τη διάσκεψη και είπε στα ξενοδοχεία όπου είχαν γίνει κρατήσεις, οι κρατήσεις αυτές να ακυρωθούν. Παρόλο που παράλληλες, τέτοιες παράλληλες διασκέψεις είναι κάτι το απόλυτα σύνηθες στη διάρκεια των συνόδων κορυφής, το Καζακστάν θεωρεί αυτή την εκδήλωση σαν μια εκδήλωση η οποία έχει σκοπό να υπονομεύσει την επίσημη σύνοδο κορυφής. Το Human Rights Watch αντιλαμβάνεται ότι δίνει προτεραιότητα ε, σε θέματα ασφάλειας στις παραμονές της συνόδου κορυφής κορυφή στην Αλλά αυτέ οι ανησυχίε δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαν αιτία για την παρεμπόδιση ή την ακύρωση των παράλληλων διασκέψεων τη κοινωνία των πολιτών. Η Human Rights Watch καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν να αποτανθεί στην ε, κυβέρνηση του Καζακστάν και να τη ζητήσει να επιτρέψει τη διεξαγωγή των παράλληλων διασκέψεων και να προωθήσει αυτή την πρωτοβουλία με κάθε δυνατό τρόπο. Ε, ε, Σα ευχαριστούμε για την τελευταία πληροφορία που μα δώσατε. Ε, εγώ έχω, τον γνωρίζω τον κύριο αυτό και έχω συνεργαστεί πολλές φορές και εξεπλάγει που μαθαίνω ότι η καζακική κυβέρνηση αντιμετωπίζει μη κυβερνητικούς οργανισμούς με αυτόν τον τρόπο ή ανθρώπους, ακτιβιστές που έχουν μεγάλη πείρα και φήμη με αυτόν τον τρόπο. Ε, υποτίθεται ότι όταν αναλάμβανε το Καζακστάν την προεδρία τη ΟΑΣΕ θα έκανε μια προσπάθεια ανοίγματο κτλ. Δεν νομίζω ότι από αυτά που μα είπατε συμβαίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, η κυρία Ζακλίν ε, Χέιλ από το Open Society Institute. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω σήμερα. Δεν θα επαναλάβω κάποιες από τις παρατηρήσεις της συναδέλφου μου για να κερδίσουμε χρόνο. Θα επικεντρωθώ μόνο σε θέματα ε, προεδρία στην ΟΑΣΕ και για το γεγονός ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα χαμένης ευκαιρίας. Οι ελπίδες που είχαμε ότι η Προεδρία της ΟΑΣΕ ε, για το Καζακστάν θα ήταν ένας καταλήτης για να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δυστυχώς ε, διαψεύστηκε. Και οι δεσμεύσει ε, που δόθηκαν το 2007 από τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών κ. Σταζίν σε κάποιο, σε πολύ, σε πολύ μέτριο βαθμό έχουν υλοποιηθεί. Ένα παράδειγμα που θέλω να σας αναφέρω είναι η ελευθερία του τύπου και η αποποινικοποίηση της συκοφαντίας. Αυτό ελπίζαμε να συμβεί, να υλοποιηθεί όταν δεσμεύτηκε στη Μαδρίτη το Καζακστάν εν ώψη της Προεδρίας του, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί και το Φεβρουάριο του 2010 δύο διάσημες ε, πλατφόρμες blog ε, θυμώθηκαν. Η κυβέρνηση ε, είχε μια υπηρεσία, δημιουργήσε μια υπηρεσία ελέγχου για να εμποδίσει την έκφραση ακραίων α, πολιτικών και θρησκευτικών. Αυτό όμως ανησυχεί πάρα πολύ την ε, κοινωνία των πολιτών της, ε, του Καζακστάν. Η συνάδελφος από το Human Rights Watch ε, ανέφερε την περίπτωση δημοσιογράφων που καταπιέζονται και καταστέλλονται και φημώνονται από την κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες. Αυτός ο δημοσιογράφος, ο οποίος πιέζεται από την κυβέρνηση, ας πούμε, επειδή υποτίθεται αποκάλυψε κρατικά μυστικά ή ένας άλλος δημοσιογράφος ο οποίος ε, έπεσε από έναν ε, ψηλό όροφο ενός κτηρίου με δεμένος πιστάγκωνα. Ε, δεν έχουν αυτές οι περιπτώσεις διερευνηθεί επαρκώς από τις αρχές του Καζακστάν. Υπάρχουν άλλα θέματα ελευθερίας πεπιθήσεων και θρησκευτική ελευθερία που συνδέονται με τα προηγούμενα. Οι πεπιθήσει αυτέ περιορίζονται παρά τους ισχυρισμού του Προέδρου ότι θέλει να είναι ανεκτική ε, η Προεδρία του και ανοιχτή. Ο νέος ε, διοικητικός ε, κώδικας και δικονομικός κώδικας προβλέπει τιμωρίες για ειρηνικές θρησκευτικές διαδηλώσεις. Μεταξύ των περιορισμών είναι λογοκρισία για θρησκευτικά θέματα, μυσαλλοδοξία από το κράτος, θρησκευτική μυσαλλοδοξία, κυρώσεις, πρόστιμα, απειλές και για καταχωρημένες και για μη καταχωρημένες θρησκευτικέ κοινότητες και άτομα. Η θρησκευτική ελευθερία δεν υπάρχει και μερικές φορές ε, γίνονται άδικες δίκες και ε, φυλακίσεις. Επίσης το έργο φιλανθρωπικών οργανώσεων περιορίζεται ε, και συχνά και, υπάρχουν και περιπτώσει όπου προσπαθεί το κράτο να βάλει το χέρι στην περιουσία θρησκευτικών κοινοτήτων. Ε, μίλησε η συναδελφό μου, μου για την συνοκορυφή τη ε, της ΟΑΣΕ στην Αστάνα. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει τότε και να μιλήσει στις αρχές ε, του Καζακστάν στην Αστάνα Υπάρχουν περιπτώσεις κακοδικίας, όπως κυρίως η περίπτωση η πιο γνωστή από αυτέ είναι του, εναντίον του Ευγέννη Ζόφτη. Επίσης τα βασανιστήρια είναι ένα τομέα όπου ελπίζουμε, ελπίζαμε και κυρίως ελπίζουμε ακόμα ότι η κυβέρνηση κάτι θα κάνει. Ε, το βασανιστήριο όμως είναι μια πρακτική πολύ συνηθισμένη και οι δράστε σε πολλές περιπτώσεις χαίρουν ατιμορρησία. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και το έχουν αναφέρει και στο παρελθόν ε, ο ειδικό απεσταλμένος της ε, ΟΑΣΕ και τον Νοέμβριο του 2009 με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το θέμα αυτό είναι πάλι ε, στο προσκήνιο σε μια συγκεκριμένη περίπτωση Ναμπούλοφ εναντίον της Ουκρανίας. Οι εκδόσεις ατόμων προς το Καζακστάν ε, είναι προβληματικές γιατί τα άτομα αυτά συχνά βασανίζονται. Τώρα, για να τελειώσω, θα ήθελα να σας πω τι ευκαιρίες έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει την ε, ευρωπαϊκή πορεία του Καζακστάν. Το Καζακστάν έχει ένα εθνικό σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε το 2009 για την τριετία 2009-2012. Αν εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο, θα υπάρξει σοβαρή βελτίωση στα ανθρώπινα δικαιώματα στο Καζακστάν. Κάνουμε έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνει τις αρχές του Καζαστάν να εφαρμόσουν το σχέδιο αυτό και να το συζητήσει στις επαφές. Ε, για τη μεταρρύθμιση κατά των βασανιστήριων. Ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση του Καζακστάν να υπάρχουν νομικές ασφαλιστικές δικλίδες ε, για την αφαίρετη σύλληψη και την ατιμορρησία των δραστών με βάση τη ε, συστάσεις τη επιτροπή του ΟΗΕ εναντίον του βασανισμού. Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφου να πιέζουν την κυβέρνηση του Καζακστάν όλοι μαζί όχι μόνο να περνάει κάποια νομοσχέδια και να προσυπογράφει διεθνείς συμφωνίες, αλλά να επιτρέπει στους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να παίζουν το ρόλο τους, να εφαρμόζει τα νομοσχέδια, τους νόμους μάλλον, να επιτρέπει και να επιτρέψει την επόμενη σύνοδο κορυφής ε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις να προσπελάσουν τη σύνοδο αυτή. Τώρα που τελειώνει η Προεδρία, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς ε, το, το Καζακστάν και το, τις προσπάθειές που κάνει ή δεν κάνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Καζακστάν θέλει να λάβει το 2012 ε, μία έδρα ε, στο Συμβούλιο για τα ανθράπινα Δικαιώματα. Θα πρέπει να διδαχθείτε εσείς από την εμπειρία σας από την Προεδρία του Καζακστάν στο ΑΣΕ και να ζητήσετε πραγματικές βελτιώσεις από το Καζακστάν ε, και πραγματική υλοποίηση των υποσχέσεών του. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Αυτά για τα θέματα της μη εφαρμογής της εφαρμογής ή μη εφαρμογής του σχεδίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την καθυστέρηση της δράσης σε ό,τι αφορά τις διασφαλίσεις σε περίπτωση αντιτρομοκρατικής δράσης. Κατά το βασανιστήριο τώρα θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Άιρμαν Κουρμάνοφ ο οποίος είναι επικεφαλής οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τάλμας είναι παρόν παρά τις τεράστιες δυσκολίες και τον προσωπικό κίνδυνο που διατρέχει για να έρθει ως εδώ. Ο Σας δίνω το λόγο λοιπόν κύριε Κουρμάνοφ. Ευχαριστώ πολύ στα ρωσικά απαντών. Κύριος Κουρμάσοφ. Είμαστε μια οργάνωση η οποία εκπροσωπεί ανεξάρτητα συνδικάτα και αντιμετωπίζουμε, αντιστεκόμαστε στις αυθαίρετες ε, συλλήψεις. Είμαστε μια οργάνωση που είναι γνωστή ως Καζακστάν 2012. Θέλω να παρουσιάσω μια αντίθετη άποψη από την επίσημη προπαγάνδα της κυβέρνησης του Καζακστάν. Το Καζακστάν κινείται υποτίθεται με μεγάλη ταχύτητα προς τη δημοκρατία και έχει υπάρξει φιλελευθερωποίηση της νομοθεσίας μας. Αλλά αυτά δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα καμία από τις υποσχέσεις που έχουν γίνει από τις εκπροσώπους της κυβέρνησης προς τον ΟΑΣΕ στη Μαδρίτη το 2007 δεν έχει εφαρμοστεί. Σε ό,τι αφορά τις ελεύθερες εκλογές, ελευθερία ε, έκφρασης, ε, ελευθερία συνεταιρίζεστε, πολιτική δραστηριότητα κτλ. Παρά το γεγονός ότι στο Σύνταγμα του Καζακστάν αναφέρεται η ελευθερία του συνέρχεστε, 90% των περιπτώσεων βλέπουν τις αρχές να αρνούνται το δικαίωμα των ε, εργατικών ενώσεων να προχωρήσουν σε διαδηλώσεις ή σε απεργίες. Όποιος αντιστέκεται, και το αντιμετώπισα εγώ τα τελευταία χρόνια, σε πολλές περιπτώσεις, δεκάδες <clears throat> ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιμετώπισαν απολύσεις. Εφέτος, επίσης, με την, ε, συνεργή, με την συνέργεια των αρχών απολύθηκαν πολλοί συνδικαλιστές λόγω της συμμετοχής τους σε νόμιμες απεργίες. Τα κράτη της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να εγγραφούν στους, και να συμμετάσχουν στις εκλογές. Κατά αυτό λοιπόν το κόμμα ΑΣΑΤ δεν θα μπορέσει να είναι παρόν στις επερχόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές. Η ελευθερία χρήσης του διαδικτύου ε, περιορίζεται δρακόντια με νομοθεσία. Οι αυτοί που διατηρούν ιστολόγια και οι δημοσιογράφοι κινδυνεύουν για αυτά τα οποία αναφέρουν. Η εφημερίδα Res Publica δεν μπορεί να τυπωθεί πουθενά λόγω απαγόρευσης από τις αρχές. Έχω εγώ αυτή την εφημερίδα η οποία τυπώνεται πια παράνομα, τυπώνεται λαθρέα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να τυπωθεί επίσημα διότι είναι πια απαγορευμένη ως ε, εφημερίδα της αντιπολίτευσης. Επίσης υπάρχει πίεση στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΤΑΝ, ο οποίος έχει, κλειστεί, έχει κλείσει από τις ε, φορολογικές αρχές. Υπάρχουν εκατοντάδες κατουμένων στο Καζακστάν που κατηγορούνται για τρομοκρατία και εξτρεμιστική δράση, ενώ βάσει των επίσημων στοιχείων δεν έχει λάβει η χώρα καμία τρομοκρατική δράση στο Καζακστάν τα πρόσφατα όλοι αυτοί που είναι <clears throat> στη φυλακή, το μόνο το οποίο έχουν διαπράξει είναι το να συμμετέχουν σε ειρηνικές Ισλαμιστικές οργανώσεις. Παραδιάζεται επίσης και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Προσφύγων. 22 Ουσπέκοι ε, πρόσφυγες έχουν συλληφθεί από τις ε, δυνάμεις ασφαλείας και θα εκδοθούν στο Καζακστάν όπου αντιμετωπίζουν θανατική ποινή. Επίσης εταιρείε οι οποίες καλλιεργούν βαμβάκι χρησιμοποιούν σε μεγάλη κλίμακα παιδική εργασία και αυτό αναφέρθηκε και από τη Human Rights Watch. Η έκθεση αυτή φυσικά δεν μπορεί να δημοσιευτεί στο Καζακτάν και η ιστοσελίδα η οποία θέλει να τη δημοσίευσει έχει μπλοκαριστεί επίσης. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτήν. Έχει περιοριστεί επίσης και η δυνατότητα εκπαίδευσης των παιδιών των οικονομικών μεταναστών που έρχονται να εργαστούν εδώ πέρα γιατί δεν έχουν το δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο. Και επίση υπάρχει περιορισμός της ελευθερίας κίνησης στο Καζακστάν σήμερα, πολύ πιο περιοριστικός περιορισμός από ό,τι ισχύει στην παλιά Σοβιετική Ένωση. Για τους κρατουμένους δεν έχει αλλάξει τίποτα σε ό,τι αφορά την απάνθρωπη μεταχείριση των κρατουμένων. Διατηρεί ουσιαστικά το παλιό σύστημα των γκουλάκ που ίσχυε στην εποχή του Σταλινισμού υπάρχουν ομάδες εσωτερικής επιβολής της τάξης στις οποίες συμμετέχουν καταδικασμένοι εγκληματίες και οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την επιβολή της τάξης μέσα στις φυλακές. Εφέτος υπήρξαν τόσες καταδιώξεις και τόσα βασανιστήρια που πολλοί ε, κρατούμενοι αυτοτραυματίζονται στην, τον Αύγουστο αυτού του έτους <clears throat> λόγω χρήσης μεθόδων από ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως παραγωγός το να βάζει κανείς τους κατουμένους να περπατούν γύρω από το στρατόπεδο ε, ακόμα και σε ακραίες συνθήκες ζέστης ή κρύου ενώ τραγουδούν τον εθνικό ύμνο του Καζακστάν έλαβε χώρα μια εξέγερση, μια μαζική λοιπόν ε, εκδήλωση όλων των κατουμένων. Σαν αποτέλεσμα ήρθαν, στείλαν το στρατό για να τους αντιμετωπίσουν, πολλοί αυτοκτόνησαν, ε, κόψανε, ε, κόψαν τις αρτηρίες τους ή ακόμα και αυτοπυρπολήθηκαν. Κανείς δεν ξέρει πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Παρά τις δηλώσεις της κυβέρνησης ότι θα εξανθρωπίσουν το σύστημα των φυλακών, τα πράγματα δείχνουν ότι όλη η πρόοδος είναι προς το χειρότερο οι οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν δημοσιεύσει σημειώματα κρατουμένων προτού χάσουν τη ζωή τους και καταδεικνύουν αυτά τα σημειώματα ότι υπάρχουν ε, εκτεταμένα βασανιστήρια στις φυλακές στο Καζακστάν χωρίς να έχει τιμωρηθεί κάποιος από το σοφρονιστικό σύστημα για αυτές τις, αυτούς βασανισμούς. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που έχουν φωνευτεί που έχουν εξαναγκαστεί σε αυτοκτονία. Όλα αυτά όμως δεν οδήγησαν σε κολασμό κάποιου από τις ε, σοφρονιστικές αρχές. Ο Κούραν είναι ένας αγωνιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πέρασε έξι χρόνια στις φυλακές για συκοφαντική δυσφήμιση. Δυστυχώς και αυτός δεν μπόρεσε να έρθει σε αυτή τη συνεδρίαση γιατί κινδυνεύει η ζωή του αλλά έχουμε την πλήρη έκθεσή του σε σχέση με την κατάσταση των φυλακών στο Καζακστάν που μπορούμε να σας δώσουμε. Έρχομαι τώρα στην πολιτική καταστολή. Στις φυλακές του Καζακστάν υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι <clears throat> όπως ο εκδότης μιας εφημερίδας ε, Σεργέποφ ο οποίος κατηγορείται για την ε, αποκάλυψη κρατικών μυστικών και ο κ. Ακάμπιαπ ο οποίος προσπάθησε να, δια, να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των εσωτερικά με, μεταναστευόντων στο Καζακστάν. Και γι' αυτό τον έχουν ρίξει στη φυλακή. Πολλές φορές αυτοί οι οποίοι διαδηλώνουν υφίστανται επιθέσεις αστυνομίας και μετά τους κατηγορούν ότι αντιστάθηκαν στη σύλληψή τους και φέρθηκαν ως χούλιγκας. υπήρξε ένα άτομο το οποίο <clears throat> καταδικάστηκε σε, δύο χρόνια φυλακής επειδή τον ξυλόδαρε ένας αστυνομικός και παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα βίντεο που καταδεικνύει ότι δεν προέβαλε καμία αντίσταση, τα δικαστήρια όμω στο Καζακστάν παρά το γεγονός ότι υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία τα αγνώρισε και προχώρησε στην καταδική και αυτά μπορούμε να σας τα δώσουμε εάν θέλετε. Και το ίδιο έγινε με τον Αρμάν Γερμίκ Μαρμίεφ, αγωνιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλακής επειδή υποτίθεται ότι επετέθη κατά της αστυνομίας και προσέβαλε ένα δικαστή. Ενώ το μόνο πράγμα που έκανε ήταν κατέβηκε σε μια διαδήλωση ζητώντας να φύγει ο πρόεδρος Ναζεμπάγεφ. Και τώρα έχει μόλις κλείσει 50 μέρες απεργίας πείνας ζητώντας από το δικαστήριο να δει το υλικό βίντεο που καταδεικνύει την αθότητά του, αλλά δεν αφήνουν κανένα σε επαφή μαζί του, ούτε τους οικείους του, είτε τους ε, δικηγόρους του. Ο Ίγκορ Κόλεφ επίση κατηγορείται για χουλιγανισμό και αυτό ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων τον, ξυλο, τον, τον δίρανε, του σπάσανε τα πλευρά του, τον έχουν ξυλοκοπήσει ιδιαίτερα, βρίσκεται κάτω από διοικητική κράτηση και η αστυνομία κάπου έχασε την καταγγελία του για Βασανισμού, και κακομεταχείριση και τον κρατήσανε για άλλες 15 μέρες για να μην φαίνονται οι μόλο, του και μετά τον στείλανε σε ένα αυτοκίνητο τον διώξανε από την <clears throat> πόλη όπου έμενε χωρίς καμία επαφή με τους οικείους του και χωρίς καμία χωρίς να του δώσουν λεφτά, χωρίς να τον αφήσουν να έχει καμία υποστήριξη. Ένας άλλος βρέθηκε στη φυλακή για 10 για 10 μέρες γιατί ήταν παρόν σε μια συνάντηση που οργάνωσε ο κύριος Χίγκινς, ο οποίος είναι εδώ ευρωβουλευτής. Υπάρχουν τρομοκρατικέ δράσει εναντίον των κομμάτων τη αντιπολίτευση των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωση των συνδικαλιστών. Όλα αυτά καλύπτονται από απόλυτη ατιμορρησία, όλε αυτέ οι επιφάσει. Ο Ταχύρ Μουχαμετζιάνοφ, συνδικαλιστή, ε, είδε το αυτοκίνητό του να ανατινάζεται. Και στη συνέχεια προσπαθήσαν να τον εγκλήσουν σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα. Και μετά από <clears throat> έρευνες οι γιατροί αρνήθηκαν να το δεχτούν και αναγκάστηκαν να τον ελαφίσουν ελεύθερο. Αλλά οι αρχές εξακολουθούν να προσπαθούν να κατασχέσουν το διαμεσμά του και έχει φυσικά ε, υποστεί ξυλοδαρμό και κινδυνεύει ακόμα. <clears throat> Είναι πολλοί λοιπόν, είναι δεκάδες οι ακτιβιστές των εργατικών ενώσεων που έχουν τύχει επιθέσεων. Δύο από αυτούς είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Και εγώ έτυχα επίθεση πριν από τη σύνοδο της, της ΟΑΣΕ πέρσι. Άγνωστοι παρέμειναν οι επιτιθέμενοι. Τα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Ουράσκ πυρπολήθηκαν και πάλι δεν βρέθηκαν ποτέ οι δράστες. Έχουν θέσει αρχές ε, ασφαλείας ναρκωτικά στις αρχές, στις στα γραφεία ε, οργανώσεων ε, αντιφρονούντων στο Καζακστάν και εξακολουθούν να εκκρεμούν διώξεις εναντίον πολλών από αυτούς τους ανθρώπους για τους ε, διαφωνούντες, ε, τους συνδικαλιστές, τους ε, ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα μέλη διαφόρων οργανώσεων. Υπάρχει μόνιμη καταστολή, παρότι το Καζακστάν έχει την προεδρία της, της ΟΑΣΕ. Υπάρχουν τόσες πολλές περιπτώσεις α, α, ΜΚΟ, ε, ειδικοί απεσταλμένοι που έρχονται εδώ για τα βασανιστήρια αλλά βλέπω νομίζω τα ανθρώπινα δικαιώματα με πολύ στενό βλέμμα και κανένας από αυτούς τους φορείς ή κανένα όργανο δεν έχει μια συστηματική ανάλυση για την επιδείνωση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν. Αν κοιτάξετε τις 50 παραγράφους του, της χάρτας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 44 από αυτές ε, Στι 44 από αυτέ ε, επιδεινώνεται η κατάσταση ε, στο Καζακστάν. Παραδείγματο χάρη, οι πολίτε δεν έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται. Είμαστε 62η σε ό,τι αφορά την στάση μας στα ΜΜΕ. Πέρυσι ήμασταν 125η με, βάση τους ε, ε, ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Τέλος, οι αρχές είπαν ότι όλοι μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές, αλλά φέτος πέρασε ένας νόμος για τον ε, ηγέτη του έθνους, όπου του δίνει η Σόβια Προεδρία ε, στον πρόεδρο Ναζαρμπάιφ και το δικαίωμα να προβάλλει βήτο ε, σε οποιονδήποτε διεκδικεί την, την αλλαγή. Αυτά. Σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας. Κύριε Κουρμάνοφ, η κυβέρνηση του Καζακστάν μας, μας έχει στείλει τον κύριο Μπεκετάια, που είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έχετε λίγα λεφτά. Έχω ένα γραπτό λόγο. Πόσο, πόση ώρα θα χρειαστείτε για να μας ε, διαβάσετε αυτό το γραπτό λόγο. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ήθελα να συστηθώ γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό και μετά θα αναφερθώ στα κύρια σημεία του γραπτού μου κειμένου. Πέντε λεπτά. Η ιστορία μου αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα που δείχνει ότι κάθε άτομο απολαμβάνει πλήρων δικαιωμάτων στο Καζακστάν. Έχει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί, να βρει μια καλή δουλειά και να εργάζεται για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Εγώ μεγάλωσα σε μια τυπική οικογένεια. Ο πατέρας μου δούλευε σε ένα γραφείο και αφού αποφύτησα από το Πανεπιστήμιο πήρα μια υποτροφία της Βρετανικής κυβέρνησης και πήγα να σπουδάσω στο London School of Economics. Στη διάρκεια της Σοβιετικής περίοδου αυτό θα ήταν κάτι το αδύνατο. Αλλά σαν αποτέλεσμα της ραγδαίας εξέλιξης στο Καζακστάν και την ανάπτυξη συνεργασίας του Καζακστάν με τον υπόλοιπο κόσμο μου δόθηκαν αυτές οι ευκαιρίες και επέστρεψα και άρχισα να εργάζομαι στο Υπουργείο Εξωτερικών μετά πήγα να δουλέψω στο γραφείο του Πρωθυπουργού, μετά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τώρα είμαι υπεύθυνο για τις μεταρρυθμίσει που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμπεριλαμβανομένων και των μεταρρυθμίσεων στο σοφρονιστικό σύστημα. Μεγάλωσα σε ένα χωριά όπου υπήρχαν ε, μάλιστα τρεις φυλακές και οι άνθρωποι από το Καζακστάν γνωρίζουν αυτό το μέρο Ζαγκριέζνη. Ο πατέρα μου δούλευε εκεί με συγχωρείτε, με σας είπα ότι έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο και έθεσαν όλοι οι προηγούμενοι μιλητές πολλά σημαντικά θέματα και θα θέλαμε να μάθουμε πώς συνεργάζεται με τους διεθνείς οργανισμούς στο Καζακστάν σε θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, αλλά θα θέλαμε να εστιαστείτε στο κυρίως θέμα δεν αγνοώ τις μεμονωμένες περιπτώσεις, τις ατομικές περιπτώσεις, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό για μένα να υπογραμμίσω ε, τις σημαντικότερες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν. Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία ε, οικουμενικής αξιολόγησης του ΟΗΕ, πάνω από 120 συστάσεις διατυπώθηκαν και δεχθήκαμε σχεδόν τις 100 από αυτές αμέσως πήραμε, μας χρειάστηκε κάποιο χρόνο για να δεχθούμε και τις υπόλοιπες, εκτός από έξι γιατί χρειαζόταν να τις μελετήσουμε περισσότερο και να αντιληφθούμε τη σκοπιμότητα τέτοιων μεταρρυθμίσεων. Από την πρώτη μέρα της μέρης της εξαρτησίας το Καζακστάν αναγνώρισε ότι ο κάθε, κάθε άτομο πρέπει να δίνει όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων του, ώστε να δημιουργηθεί ένα κοσμικό ε, δικαιοκρατικό καθεστώς στη χώρα βασανιστήρια δεχθήκαμε έναν ειδικό εισηγητή, τον Μάνφρεντ Νόουακ, για τα βασανιστήρια και του ζητήσαμε να επανέλθει. Είπε ο ίδιος ότι το Καζακστάν είναι η μόνη χώρα η οποία καλεί ε, ειδικό εισηγητή για νέα επίσκεψη παρακολούθησης για να διαπιστώσει τι ολοκληρώθηκε και τι βρίσκεται υπό εξέλιξη. Ε, πρόκειται να καθιερώσουμε μηχανισμούς που θα εμποδίζουν, θα, δεν θα επιτρέπουν τα βασανιστήρια σε χώρους κράτησης. Πρόκειται να αποποινικοποιήσουμε 36 ε, ε, εγκλήματα ή αδικήματα με μεταρρύθμιση του ποινικού μας κώδικα. Σχεδιάζουμε επίσης να καθιερώσουμε νέες μορφές κυρώσεων και ποινών που δεν θα ε, περιλαμβάνουν την κράτηση, τη φυλάκιση για διάφορες περιπτώσεις. Το Καζακστάν είναι ανοιχτό σε οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας συνεργαζόμαστε επικοδομητικά με πολλούς διεθνείς οργανισμούς σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση του σοφρονιστικού συστήματος και του ποινικού μα δικαίου. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά με τον Μάνφρεντ Νόλ, τον οποίο συνάντησε εγώ στη διάρκεια του έργου του τέσσερις φορέ. Σαν χώρα λοιπόν το Καζακστάν ανοιχτή, είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε συνεργασία και καλούμε όποιον ενδιαφέρεται να έρθει να επισκεφθεί το Καζακστάν. Πολλέ από τις υποθέσεις που αναφέρθηκαν από τους εκπροσώπους των ΜΚΟ από τον εκπρόσωπο των ΜΚΟ έχω άφθονο υλικό για όλες αυτές τις υποθέσεις και είμαι έτοιμος να τον συναντήσω απόψε αργότερα και να τα συζητήσουμε όλα λεπτομερώς. Αν κάτι δεν συζητηθεί εδώ, είμαι διατεθειμένος να δεχθώ οποιονδήποτε στη χώρα για να το συζητήσουμε. Επειδή δεν υπάρχει χρόνος θα σταματήσω εδώ και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα δείγμα συνεργασίας. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας θέσω ένα ερώτημα για την διάσκεψη των μη κυβερνητικών οργανώσεων που θα γινόταν υποτίθεται παράλληλα με τη Σύνοδο Κορυφής της ΟΑΣΕ στην Αστάνα. Νομίζω 1 και 2 Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρός σας θα συναντήσει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αύριο και καλό θα ήταν να ακούσουμε εν ώψη αυτής της συζήτησης εάν θα επιτρέψετε την διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Όλο το απόγευμα συζητάμε πολύ σοβαρά με την κοινωνία των πολιτών, με τις οργανώσεις που μας ενημερώνουν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συνεργαστείτε με την ε, κοινωνία των πολιτών. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι δυνατόν να παραμελείτε με τέτοιο τρόπο τη χάρτα του Ελσίνκη. Όλοι οι ανθρώπινοι, το θέμα των, ε, της ανθρώπινης συνεργασίας, ανθρώπινης διάστασης, ε, είναι η συνεργασία. Γνωρίζω αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι υπάρχει παρεξήγηση όλα τα ξενοδοχεία στην Αστάνα, γιατί η Αστάνα δεν είναι πολύ μεγάλη πόλη, όλα τα ξενοδοχεία έχουν γεμίσει ήδη, έχουν γίνει κρατήσεις από τον Αύγουστο για αυτά. Είμαι σε, ήμουν σε μια συνάντηση όπου συζητήθηκε αυτό το πρόβλημα και αποφασίστηκε ότι οι τοπικές αρχές στην Αστάνα θα βοηθήσουν τους διοργανωτές να βρουν ένα χώρο να, για να διεξαχθεί το συνεδριό τους. Δυστυχώς όμως θα δυσκολευτούν να βρουν δωμάτια εκείνες τις ε, ημερομηνίες. Αλλά όμως γίνεται μια προσπάθεια να τους βοηθήσουν να βρουν δωμάτια. Όμως οι τοπικές αρχές θα ασχοληθούν με το θέμα αυτό και δεν υπάρχει καμία εντολή, καμία δράση για να σταματήσουν αυτή την την παράλληλη εξαγωγή της, του συνεδρίου. Κυρία Αντριάννα Μπέργκ, ποια είναι η δική σας εντύπωση. Από, τι ό,τι γνωρίζω, εγώ μίλησα με μερικούς από τους οργανωτές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΟΑΣΕ στην ε, Βασοβία. Είχαν ε, πληρώσει για μια αίθουσα συνεδρίασης και 17 δωμάτια και τελικά ακυρώθηκαν σε αυτές οι κρατήσεις. Και κλείνει το μικρόφωνο της κυρία Αντριάννα. Ναι, νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε να συζητούμε αυτό το συγκεκριμένο θέμα γιατί είναι κατεπίγον. Είναι μονάχα ένα μήνα που μα χωρίζει από αυτό το γεγονό. Χωρί μικρόφωνο. Μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο. Επίση, υπάρχει πληροφορία ότι την 1η και 2η Δεκεμβρίου θα κλείσει το αεροδρόμιο τη Αστάνα για λόγου ασφαλεία. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες στην ε, συνεδρία σε αυτή την παράλληλη δεν θα μπορούν να φύγουν από την Αστάνα κάτι διάρκεια αυτών των ημερών. Ο τελευταίος μας ομιλητής, εφόσον δεν ζητάει κανείς άλλο το λόγο, είναι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, ο υπεύθυνος της Μονάδος για την Κεντρική Ασία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομος θα είμαι, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο και θα εστιάσω κυρίως ε, στην Προεδρία της ΟΑΣΕ και τα σχετικά θέματα. Είμαστε απογοητευμένοι, μπορούμε να το πούμε αυτό, για τον τρόπο με, το τον οποίο το Καζακστάν υλοποίησε τις δεσμεύσεις και τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις που έκανε κατά την ε, προσπάθεια και εκστρατεία να αναλάβει την ε, Προεδρία της ΟΑΣΕ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από το Καζακστάν και να προχωρήσουν οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Οι αλλαγές που έχουν γίνει από το Κοινοβούλιο στο Καζακστάν για τους νόμους, για τις εκλογές, για την, ε, τα πολιτικά κόμματα, την ε, αυτοδιοίκηση, δεν έχουν γίνει σεβαστοί. Ο αριθμός των μελών για να γίνει δεκτό ένα καινούριο κόμμα έχει μειωθεί από 50.000 σε 40.000 μέλη, αλλά είναι πολύ μεγάλο αυτό το νούμερο για να ενθαρρύνουμε οποιονδήποτε να ασχοληθεί με την πολιτική για να προωθήσουμε α, τον πολιτικό πλουραλισμό το 7%. 7% το όριο για να μπει κανείς στο κοινοβούλιο είναι υπερβολικά ψηλό. Υπάρχει ένας μηχανισμός που έχει δημιουργηθεί για να επιτρέψει και σε ένα δεύτερο κόμμα να μπει στο κοινοβούλιο. Ακόμη και αν δεν πάρει το 7% των ψήφων. Νομίζουμε ότι στην πραγματικότητα οι αλλαγές αυτές είναι μικρές για το νομοσχέδιο για, το, για τα ΜΜΕ και υπάρχει ακόμα ε, το πρόβλημα με την α, δυσφήμιση που παραμένει ποινικό αδίκημα. Ε, με βάση το δίκαιο του Καζακστάν υπάρχουν έξι άρθρα ε, που προστατεύουν την τιμή των πολιτικών αξιωματούχων, ιδίως του Προέδρου. Μας ανησυχεί αυτό και μας ανησυχούν οι επαναλαμβανόμενες δίκες ε, εναντίον ανεξάρτητων ε, εφημερίδων ε, που τους περιορίζει τη δυνατότητα λειτουργίας τους. Και το γεγονός ότι η θέση σε ισχύ μιας περιοριστικής νομοθεσίας για το ίντερνετ δεν βοηθάει την ελεύθερη έκφραση. Το, τέλος, για το νομοσχέδιο για την αυτοδιάθεση οι αλλαγές που έχει εισαγάγει το Κοινοβούλιο δεν νομίζουμε ότι αποτελούν πραγματική βάση για πραγματική αυτοδιοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαστε απογοητευμένοι από την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έκανε το Καζακστάν. Ένα άλλο θέμα, το θέμα της έγκρισης του νομοσχεδίου ε, για τον ηγέτη του έθνους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούσαμε τα άκουσε τα επιχειρήματα του Προέδρου Ναζάρ Μπαϊεφ που δικαιολογούν δικαιολογεί ας πούμε την άρνηση της υπογραφής του νομοσχεδίου. Παρ' όλα αυτά όμως ετέθησε ισχύ το νομοσχέδιο. Αυτό μας εξέπληξε βέβαια. Επίσης πολλά πολλές στοιχείες της νέας νομοθεσίας δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις και τις ε, αξίες της ΟΑΣΕ. Και πιστεύουμε ότι δεν βοηθούν την πορεία εκδημοκρατισμού της χώρας αυτής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ όλες τις πλευρές για όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώσαμε στη διάρκεια αυτής της σύντομης ακρόασης. Έχω ένα συγκεκριμένο μήνυμα που θα ήθελα να μεταφέρω στους φίλους μας από το Καζακστάν είναι από το γραφείο του Προέδρου Μπούζεκ και είναι το εξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσβλέπει σε αυτή την ανοιχτή ανταλλαγή που προσφέρει το Καζακστάν και αύριο στη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Μπούζεκ. Η συζήτηση λοιπόν θα συνεχιστεί και θα παραμείνουμε σε επαφή με τον κύριο Κουρμάνοφ και αναμένουμε ότι δεν θα υπάρξουν αντίπεινα ή οτιδήποτε τέτοιο διότι ακούσαμε πολλά ανησυχητικά παραδείγματα για το τι παθαίνει κανείς όταν εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στον Καζακστάν. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτή η παράλληλη διάσκεψη ή συνάντηση τη κοινωνίας των πολιτών θα μπορέσει τελικά να λάβει χώρα, διότι θα είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη εκδήλωση στη διάρκεια της οποίας θα μπορέσει να γίνει μια συζήτηση για το πώς μπορεί να αναπτύξει και να ενισχύσει την προσέγγιση του στα ανθρώπινα δικαιώματα ο ΟΑΣΕ. Ευχαριστώ.